Buongiorno. Ieri sera si è riunito il gruppo dei coordinatori. Λοιπόν, οι συντονιστέ δεν αποφάσισαν και πάρα πολλά πράγματα. Τέθηκε το θέμα του Ουγγρικού Συντάγματο και είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε το έγγραφο της ομάδας της Βενετίας έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να το μελετήσουμε πολύ προσεκτικά, συγκριτικά θα έλεγα το θέμα. Να Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω όμως είναι ότι σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το συζητήσαμε γιατί σήμερα το απόγευμα υπάρχει στο Παρίσι μια διακοινοβουλευτική συνάντηση και εμείς υποστηρίζουμε ότι στα πλαίσια των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν να υπάρξει μια γραπτή συμφωνία και η υποψηφιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποψηφιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δικαστήριο του Στρασβούργου να προωθηθεί σύμφωνα με το 156 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ένωσης, δηλαδή από την ομάδα η οποία επιλέγει ήδη τους υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αποφασίσαμε επίσης η τακτική συνάντηση που προβλέπεται για την 4η Οκτωβρίου να μεταφετεθεί στην 5η, στην 4η μάλλον 5 Οκτωβρίου. Προφανώς εννοούσε τρίτη ο Πρόεδρος. Ένα άλλο θέμα αφορά ένα έγγραφο της Επιτροπής Αναφορών. Διεκδικεί η οκτωβριου να μεταφερθεί στην 5 η στην 4 η μαλλον 5 οκτωβριου προφανως εννοουσε τριτη αυτή να θεωρηθεί αρμόδια επί της ουσίας για την οργάνωση ακροάσεων μετά από τη συλλογή ε, των υπογραφών για μια πρωτοβουλία των πολιτών, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη. Εμείς είπαμε ότι το θέμα των αναφορών είναι διαφορετικό από την πρωτοβουλία των πολιτών και πρέπει να εμείνουμε στην κανονική διαδικασία. Συνεπώς λοιπόν η αρμοδιότητα της Επιτροπής Αναφορών είναι συζητήσιμη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλο θέμα είναι οι αναφορές, άλλο θέμα η πρωτοβουλία των πολιτών. Εν πάση περιπτώσει θα στείλουμε μια επιστολή διευκρινίζοντας ε, την πλευρά αυτή γιατί θεωρούμε ότι και εμείς είμαστε αρμόδιοι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά που συζητήσαμε χθες το απόγευμα σε επίπεδο συντονιστών. Μπορούμε νομίζω να ξεκινήσουμε την κανονική μας συνεδρίαση. διευκρινίζοντας, γιατί είναι υποχρεωτικό αν και το ακούτε συνέχεια, ότι υπάρχει αναμετάδοσή μας διαδικτυακή των συνεδριάσεών μας. Θα συζητήσουμε την έκθεση Μάρτιν σε αυτή τη φάση, η οποία έμεινα από χθε και αφορά το δικαίωμα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μάρτιν, ο οποίος θα μας πει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε και θα γίνει μια πρώτη συζήτηση αμέσως μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που φέρετε το θέμα μπροστά. Γνωρίζουμε, συνάδελφοι, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το, το δικαίωμα να θεσπίσει προσωρινές επιτροπές για να εξετάζει υποτιθέμενα προβλήματα κακοδιαχείρισης. Πράγμα το οποίο αφορά όχι μόνο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα κράτη-μέλη και τα σχετικά τους όργανα. Θέλω αυτό να το υπογραμμίσω, διότι είχαμε κάποιες αμφιβολίες ακούσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Έχουμε φέρει πριν θεσπίσει προσωρινή επιτροπή για την εξέταση των έκτακτων παραδόσεων των, ε, με βάση τον κανόνα, το άρθρο 145-146 του κανονισμού. Ε, αλλά αυτές είναι οι προσωρινές. Οι εξεταστικές επιτροπές έχουν να κάνουν με κακοδιαχείριση ή εσφαλμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Και έτσι έχει το δικαίωμα το Κοινοβούλιο να θεσπίσετε είδους εξεταστικές επιτροπές και να διεκδικήσει και στους εξουσίες του Κοινοβουλίου με την άσκηση αυτών των ε, ανακρατικών διαδικασιών. Από το 1995 μόνο τρεις φορές έχουν θεσπιστεί τέτοιες επιτροπές. Δεν είναι καθημερινό δηλαδή ε, φαινόμενο. Ούτε καν εμφανίζονται άπαξ, ε, έστω. Δεν εμφανίζονται πάντοτε σε κάποια θητεία κοινοβουλευτική. Είχαμε όμως εξεταστικές για το καθώς τη μετακόμισης, για τη σπογγόδια κεφαλοπάθεια και για την ε, Equal Life, για την ασφαλιστική. Την έκθεσή μου την εμπνέομαι λίγο πολύ από την υπόθεση της Equal Life, της ασφαλιστικής, γιατί ακριβώς ε, απεδείχθη από αυτή την ε, περίπτωση ότι δεν υπήρχαν επαρκείς εξουσίες ώστε να μπορέσει, δεν προβλέπονταν αρκετέ εξουσίε ώστε να μπορέσει να τελέσει το έργο τη αυτή η Εξεταστική Επιτροπή και να διερευνήσει την υπόθεση. Η συνθήκη δεν προσδιορίζει συγκεκριμένου όρου άσκηση αυτή τη ανακριτική διακριτικότητα τη Εξεταστική Επιτροπή. Μόνο προβλέπει τη δυνατότητα εξέταση μια υποθέσεω μέσω μια Εξεταστική Επιτροπή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να θεσπιστούν στην πράξη αυτές οι αρμοδιότητες και στη συνέχεια έχουμε το άρθρο 226 όπου λέει ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Δία Πρωτοβουλία σε διαλλαγή, σε συνεννόηση με το, με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσει και να προσδιορίσει τους όρους λειτουργίας μες της Εξεταστικής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν προτείνουμε να ε, αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας γιατί είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά που έχουμε τη δυνατότητα για άσκηση τέτοιων ε, εξουσιών. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι πορίσματα προκύπτουν από την Equalife. Καταρχάς ότι δεν υπάρχουν ε, εξουσίες, δεν υπήρχαν μάλλον εξουσίες ως προς, το, τη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ε, διερευνήσει μια υπόθεση παρά μόνο στο να καταγγείλει κάποια που θεωρούσε υπέτειο για κακοδιαχείριση. Δηλαδή μπορούσαμε ακόμη και να έχουμε καλέσει μάρτυρες και αυτοί να αρνηθούν να προσέλθουν να μιλήσουν. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε οποιαδήποτε κύρωση ή δεν υπήρχε η κύρωση σε περίπτωση ψευδομαρτυρίας. Δεν υπήρχε δυνατότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κληθούν μάρτυρες μέσω των εθνικών δικαστηρίων. ούτε να επιλέξουμε ποιον θέλουμε να ακούσουμε. Μόνο ε, όταν απευθυνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο φορέα ή οργανισμό, η διοίκηση του εν λόγω φορέα αποφάζει ποιον θα μα στείλει για να μα μιλήσει. Αλλά δεν μπορούμε να στήσουμε συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν και χωρίς βέβαια να διεκδικούμε μια λευκό επιταγή η οποία θα μας επέτρεπε να ανοίγουμε οποιοδήποτε τα σιρτάρια και τα τουλάπια και να ζητούμε οποιοδήποτε να έρθει ενώπιον μας, ζητούμε στην πρόταση αυτή θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη-μέλη, φυσικά πρόσωπα, να μπορούν να κληθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των, της εξεταστικής αυτής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να δώσουν απαντήσεις ε, ακριβείς και αληθείς στις ερωτήσεις που θα τους τεθούν. Λέω επίσης ότι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας χορηγήσει πληροφορίες και θα πρέπει η Επιτροπή καταρχάς να μπορεί εκείνη να αποφασίσει ποιον θα μας στείλει, αλλά εάν στη διάρκεια αυτή τη διαδικασία εμεί διαπιστώσουμε ότι κάποιος συγκεκριμένος κάποιο φυσικό πρόσωπο δηλαδή που υπάρχει στην Επιτροπή γνωρίζει πράγματα που θέλουμε να ε, ακούσουμε, τότε θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κλητεύσουμε τον εν λόγω άνθρωπο. και χωρίς να θέλω να υπερβάλλω ε, της, ε, τον αντίκτυπο αυτής της ρύθμισης, πιστεύω ότι θα υπάρχει δυνατότητα για τους λεγόμενους whistleblowers, εκείνους δηλαδή που καταγγέλουν ε, τα κακό κείμενα, να μιλήσουν πιο ανοιχτά και πιο ελεύθερα ενώπιόν μας, χωρίς να φοβούνται. Και έτσι προχωρώ στην επόμενη σύσταση, όπου ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να υποτάσσονται σε τέτοια αιτήματα. Με βάση τον ε, κανονισμό δηλαδή θα πρέπει να ε, αναπτυχθεί αυτό το επίπεδο συνεργασίας. Οι κυρώσεις θα έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε διαγνωστή απαραβίαση, παράβαση μάλλον άρνηση για προσέλευση μάρτυρα, ψευδορκία, και ούτω καθεξής. Η Εξεταστική Επιτροπή θα συλλέγει στοιχεία, πραγματικά και περιστατικά, με στόχο να διευκρινίσει τι έχει συμβεί και πότε. Άρνηση συνεργασία θα συνεπάγεται κυρώσει. Ω προ του ιδιώτε, τα κράτη-μέλη θα αναλαμβάνουν με βάση το εθνικό του δίκαιο ε, τη σχετική δράση και για να είναι οι κυρώσει ισοδύναμες δίκες ε, τροποντινά θα πρέπει να αναλαμβάνουν ε, δράση και σε περίπτωση σπάνια μη συμμόρφωσης και υπαλλήλων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων με κύριο επιχείρημα σε όλα αυτά να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον της κοινότητας. Δεν υπάρχει ε, περίπτωση να παραβλαφθεί το συμφέρον της, τα συμφέροντα της κοινότητας. Αντιθέτως θέλουμε να διερευνούμε οποιαδήποτε προβλήματα τέτοια ακριβώς για να προλαβαίνουμε και να προφυλάσσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης σημειώνω ότι δεν υπάρχει δεδομένο πόρισμα μια τέτοια επιτροπής η ετοιμιγορία της μπορεί να έχει να κάνει και με την συνέχιση της εξέτασης, την παραπομπή σε άλλους φορείς ή θεσμικά όργανα, η Εξαστική αυτή Επιτροπή έχει σαν ρόλο να αναζητήσει την αλήθεια. Και αυτό θα πρέπει να μπορέσει να πράξει. Και επαναλαμβάνω, οι κυρώσεις μας, οι κυρώσεις οι αναφέρομαι έχουν να κάνουν όχι με την επιβολή κάποιας τιμωρίας που θα απορρέει από τα ευρήματα αυτής της Επιτροπής, αλλά μόνο με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που κάποιο δεν συνεργάζεται μαζί μα, δηλαδή δεν προσέρχεται ο μάρτυρα, ψευδορκή και ούτω Εάν από το πόρισμα των εργασιών αυτή τη Επιτροπή προκύψει κάποια κλιματική ενέργεια, αποδειχθεί κάποια κλιματική ενέργεια, αυτή θα πρέπει να τιμωρηθεί με βάση τι διατάξει που ισχύουν αλλαχού. Ευχαριστώ. Κάποια στιγμή ήμουν αφηρημένος. Θα ήθελα όμως να μάθω κύριε Μάρτιν οι τρεις προηγούμενες επιτροπές έρευνας, τις οποίες εσείς αναφερθήκατε, ποιες είναι, δεν το κατάλαβα καλά. Με ακούτε. Ναι, Πρόεδρε. Ήταν η... το καθεστώς διαμετακόμισης, το κοινοτικό καθεστώς διαμετακόμισης, ε, επιδοτήσεις δηλαδή της ΚΑΠ και άλλα θέματα πάνω από όλα που είχαν να κάνουν με την ε, κινητικότητα γεωργικών προϊόντων που είχαν επιδοτηθεί ήταν η σποκώδηση κεφαλοπάθεια και η Equal Life που οδήγησε σε ανάληψη δράση από την ε, καινούρια κυβέρνηση της Βρετανίας αλλά η προηγούμενη ξέρετε δεν είχε αναλάβει δράση και σε ήταν της μου κομματικής Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτιν. Νομίζω ότι το δικαίωμα έρευνας είναι αναπόσπαστο τμήμα των εποπτικών αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου αναζητεί την αλήθεια για θέματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. θα έπρεπε να μπορεί να λειτουργήσει σε κάποιες περιπτώσεις και σαν δικαστήριο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, απλά καλύπτουμε κάποια κενά και εδώ θα πρέπει να καλύψουμε και την περίπτωση της κακής κακοδιοίκησης γενικά των κοινοτικών οργάνων. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα όργανα και να έχουμε δικαίωμα να συλλέγουμε όλα τα έγγραφα τα οποία άπτονται της συγκεκριμένης κακοδιοίκησης. <clears throat> θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παίρνουμε πληροφορίες και από την Ένωση και από τα εθνικά όργανα και από νομικά πρόσωπα και από φυσικά πρόσωπα. Οι επιτροπές έρευνας θα πρέπει να είναι σε θέση να καλούν ε, πολίτες της Ένωσης, δημοσίους υπαλλήλους, ε, ε, έμπειρους γενικά σε κάποια θέματα έτσι ώστε να μπορούμε να ερευνούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την συγκεκριμένη περίπτωση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί η πρόταση του κυρίου Μάρτιν είναι μια καλή βάση για περαιτέρω συζητήσεις. Ο κύριος Άγνιου. Thank you, Chairman. Uh, uh, I'd ευχαριστώ ήθελα να πιστήσω την ε, προσοχή της Επιτροπής στην, ε, παρά... στην σελίδα 6 όπου αναφέρεται το κλητεύονται και ε, αναδιρωτώ με κατά πόσο υπάρχουν κάποια λάθη στην αγγλική μετάφραση γιατί υπάρχουν κάποια άλλα σφάλματα. Ο κύριος Μάρτιν χρησιμοποιεί αυτό τον όρο δύο ή τρεις φορές στο κείμενό του και νομίζω ότι αυτή είναι μια ζωφερή εξέλιξη γιατί το να κλητεύονται αυτό συνεπάγεται μια βία ε, δεν ξέρω, δεν ε, υπήρξε καμία επιλογή μέσω της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Ε, θεωρείται ότι κάποιος, σε κάποιον ασκείται βία και προσαγάγεται βία στο, στην ακρόαση, στην, να καταθέσει μια μαρτυρία. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι δεδειγμένη χρήση βίας. Το άλλο θέμα το οποίο θέτει είναι το whistleblowers και νομίζω ότι εδώ ίσως υπάρχει κάποια υποκρισία. Ε, νομίζω επενθυμίζει τις ε, βρετανικές ε, απικίες. Μπρόνς, ευχαριστώ. Όπως ε, υπόθηκε η προτινόμενη νομοθεσία θα ενισχύσει την υποχρεωτική παρουσία των προσώπων όχι μόνο θα την επιβάλλει, αλλά θα επιβάλλει επίσης και την υποχρέωση απάντησης στις ερωτήσεις. Αυτό είναι μια παρέμβαση στην προσωπική ζωή των πολιτών. Εγώ δεν λέγω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ποτέ δικαιολογημένο ή θεμητό, αλλά θα είναι δυνατόν για τα δικαστήρια των κρατών να επιβάλλουν την παρουσία και την υποχρέωση απάντησης. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όμως ακόμα ένα κυρίαρχο κράτος, αν και έχει βέβαια φιλοδοξίες να γίνει. Να ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Οι εξουσίες αυτές ξεπερνούν τις εξουσίες των ειδικών επιτροπών της Κάτω Βουλής. Οι επιτροπές της Κάτω Βουλής μπορούν να καλέσουν μάρτυρες. Αν δεν παραστούν οι μάρτυρες τότε μπορεί να διωχθούν για περιφρόνηση προς το Κοινοβούλιο. Ε, θυμάμαι την περίπτωση της Εντουίνα Κάρι όπου είχε κληθεί σε μια τέτοια συνεδρίωση και σε άλλες περιπτώσεις ήλθαν εκεί αλλά δεν έδωσαν τις κατάλληλες απαντήσεις βέβαια. Εν πάση περιπτώσει οι αρμοδιότητες αυτές δεν θα πρέπει να δοθούν σε ένα υπερεθνικό σώμα όταν μερικές φορές δεν υπάρχουν οι αρμοδιότητες αυτές ακόμα και στις αρμόδιες επιτροπές των κοινοβουλίων των κυρίαρχων κατά τα άλλα κρατών. Ο κύριος Νταφ. Θεωρώ θετικό το ότι ξεκινά εκ νέου η εξέταση αυτού του δικαιώματος πρωτοβουλίας που μας χορηγεί η συνθήκη της Λισαβόνας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. <clears throat> Νομίζω ότι το δικαίωμα στη διεξαγωγή μιας ερευνητικής διαδικασίας όπως επίσης και το δικαίωμα θέσεως ερωτήσεων είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό ενός κοινοβουλίου. Και υπάρχει φυσικά, με διαφορετικές βέβαια μορφές, το δέχομαι αυτό, αλλά υπάρχει σε όλα τα κοινοβούλια. Ιστορικά είναι αρκετά περίεργο βέβαια το κοινοβούλιο μας να έχει χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα μόνο σε τρεις περιπτώσεις. Θα προέβλεπα μια πιο τακτική προσφυγή στην δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας μετά από την θέσπιση αυτού του νέου νομοθετικού μέτρου. Έχει σημασία λοιπόν να θεσπιστεί σωστά. Φυσικά και δεν είμαστε δικαστήριο, αλλά είμαστε ή μη δικαστικό ή σχεδόν δικαστικό ε, στον τύπο τουλάχιστον σώμα. Γνωρίζουμε επίσης ποιες είναι οι διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες οι οποίες υπάρχουν εδώ και θα πρέπει φυσικά να τις λάβουμε υπόψη μας με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Μάρτιν. Πρώτον, τι γίνεται με τον Ombudsman δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η διαδικασία της Επιτροπής Έρευνας και σε ποιο βαθμό είναι συμβατή η βελτίωση αυτή με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει ο Ombudsman για να αποδέχεται παράπονα για κακοδιοικήσεις κτλ. Θα ήθελα να μου πει λοιπόν ο David Μάρτιν αν έχει συζητήσει με τον Ombudsman για την διαδραστικότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις ε, έρευνες του Κοινοβουλίου και τις αντίστοιχες του Ombudsman. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εδώ ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνουμε στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες του Ombudsman, του διαμεσολαβητή και θα πρέπει επίσης να καλείται ο διαμεσολαβητής να συμπαρίσταται, να έρχεται αρρωγός στις ε, έρευνες τις οποίες κάνει το Κοινοβούλιο, χωρίς όμως όπως είπα να φύγονται ε, τα στοιχεία αυτονομίας ενός διαμεσολαβητή. Το δεύτερο θέμα είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω ακόμα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς οι οποίοι αρνούνται να καταθέσουν αφού κληθούν. Ιδιαίτερα δημόσιους υπαλλήλους κρατών μελών. Τώρα αυτά που λέω πιθανολογώ ουσιαστικά, αλλά υποπτεύομαι ότι θα μπορούσε ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι πολύ συχνά να καλούνται να δώσουν εξηγήσει για τις πιθανές παραβιάσεις των χρηστών πρακτικών στα πλαίσια της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει συνταγματικές συγκρούσεις θα έλεγα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν υπάρξει αρκετές τέτοιες συγκρούσεις και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να προσθέσουμε επιπλέον. Στη σελίδα 17, παράγραφος 43, μάλλον άρθρο 43, σχετικά με την ορκομοσία, με τον όρκο μάλλον. Όταν έχω πάει στα δικαστήρια μου ζητούν να ορκιστώ πριν δώσω την κατάθεση και όχι μετά φυσικά την κατάθεσή μου. Και είναι λίγο περίεργο η διατύπωση εδώ στα αγγλικά είναι κάτι το οποίο ίσως να μην είναι πολύ κατανοητό. That formulation ε, ε, ε, comes from. And Κάτι τώρα σχετικό με το χρονοδιάγραμμα. Πότε πιστεύετε εσείς ότι μπορούμε να προωθήσουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Πιστεύετε ότι η Πολωνική Προεδρία είναι διατεθειμένη να αναλάβει να το προωθήσει. Η κυρία Γιέτερ Μάκη. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, Οι Βρετανοί συνάδελφοι ε, ανησυχούν όσον αφορά την έννοια το λέξη σάμοντ, ε, κλητεύονται ή καλούνται οι μάρταρες. Αλλά θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στις εποπτικές εξουσίες. Θεωρώ ότι είναι βέβαιο ότι όλες οι χώρες μέλη ενδιαφέρονται να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν ενδιαφέρονται ε, δυστυχώς για το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες ή στις ίδιες τους χώρες, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτές τις εποπτικές εξουσίες, αρμοδιότητες και νομίζω ότι όλες οι χώρες μέλη και οι εθνικές κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για το πώς χρησιμοποιούνται ε, τα χρήματα, για παράδειγμα, τα κονδύλια της αναπτυξιακής βοήθειας και μεταβαίνουν προς διάφορες χώρες και προσπαθούν να εξετάσουν περιπτώσεις ενδεχόμενης κακοδίκησης. Αυτό ίσως ε, είναι ένα θέμα. Εγώ δεν είμαι φεντεραλίστρια, αλλά θεωρώ ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια χρήματα θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακολουθεί, να υποπτεύει το πώς χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η διοίκηση λειτουργεί καλά. Είναι το καθήκον μας. Ah, Πριν να... Α, κάποιος ο κύριος Άγνιο έχει δει ξανά το λόγο. Ναι, πρόεδρε. Θα επανέλθω σε αυτό. Ε, τι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δόθηκαν στην περίπτωση της Equitable Life, του σκανδάλου αυτού. Δεν έχουν ε, ζητήσει άλλοι το λόγο και θα κλείσει τη συζήτηση ο συνάδελφος Μάτιν. Θα ήθελα να θέσω κι εγώ μια ερώτηση. Πιστεύω ότι σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες προβλέπεται το κοινοβούλιο τους να μπορεί να διεξάγει κάποιες έρευνες. Μια συγκριτική μελέτη αυτών τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο κρατών μελών θα είχε ενδιαφέρον. Υπάρχει μια κάποια τέτοια μελέτη. Μια παρατήρηση επίσης Στην Ιταλία έχουμε κάνει πάρα πολλές ερευνητικές επιτροπές για θέματα διαφθοράς κτλ. Και το θέμα το οποίο τίθεται είναι το των σχέσεων με την δικαστική εξουσία. Ε, στρεβλώσεις, ε, γενικά αδικαιολόγητες πιέσεις και τα λοιπά, πολιτικές ή όχι. Στην περίπτωσή μας λέγεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια έρευνα αν διεξάγεται μια δικαστική έρευνα και ε, προβλέπεται ότι αν ξεκινήσει μια δικαστική έρευνα μετά την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον χρόνο διάρκειας της δικαστικής διαδικασίας διακόπτεται η κοινοβουλευτική. Δεν θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή Έρευνας να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και τους ίδιους ρόλους με ένα δικαστικό σώμα. Τα δικαστικά σώματα είτε διαπιστώνουν ή δεν διαπιστώνουν την ύπαρξη ε, πλημελημάτων, κακουριμάτων κτλ. ή τον σεβασμό ή όχι των δικαιωμάτων των ε, εμπλεκομένων. Εμείς δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Εμείς έχουμε αρμοδιότητες πολιτικές, έχουμε αρμοδιότητες διαπίστωσης της χρηστής ημί διοίκησης, δεν έχουμε δυνατότητες επιβολής ποινών κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αποφύγουμε οι δικαστικές έρευνες να δημιουργούν προβλήματα στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Δεν ξέρω τι λύσεις μπορεί να βρεθούν, είναι σαφές πάντως ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ουσιαστικά ε, υπεράνω των δικαστικών αρμοδιοτήτων. Πάντως θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε αυτό που είπα προηγουμένως για το τι πράγματι ισχύει στα διάφορα κράτη-μέλη με τα... να κάνουμε μια σύγκριση. Κύριος Μάρτιν. Thank you very much, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις καλές και σημαντικές ερωτήσεις. Για την κυρία Γιάτσαρμακή. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Προφανώς είμαστε στο ίδιο μήκος αν έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ε, για τροποποίηση του κειμένου, δεδομένου ότι ξεκινάμε από την ίδια βάση, ότι δηλαδή εφόσον έχουμε μια εξαστική επιτροπή σε ένα κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση αυτή να καλεί μάρτυρες και να εξετάζει αποδεικτικά για να καταλήξει σε μια ε, σε ένα πόρισμα, σε μια εκδοχή του τι έχει συμβεί. Πριν επανέλθω για τα υπόλοιπα θα απαντήσω στο ερώτημα της Equal Life ότι δεν μιλούμε μόνο για ε, παραβίαση ή για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχουμε να κάνουμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και άλλωστε τα παιδέχθη ίδια η Βρετανική κυβέρνηση, με μη εφαρμογή οδηγιών που έπρεπε να ισχύουν στο Βρετανικό δίκαιο. Και εξαιτία αυτών εθίγησαν οι παθόντες, οι οποίοι ήταν εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες και θα θυμάστε όσοι ήσασταν τουλάχιστον εδώ την εποχή αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ερχόντουσαν ε, πολλοί άριθμοι παθόντες να μιλήσουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Για τον κύριο Άντνιου λυπούμε που βλέπει τα πράγματα, την ειδικόνα αυτή της κλίσης μάρτυρα ως ζωφερής εξέλιξης. Είναι ο κατάλληλος τρόπος αυτός. Έχουμε το δικαίωμα να καλέσουμε μάρτυρα Απλώς πιστεύω και δεν θα θέλει ασφαλώς και ο κύριος Σάββιν με τέτοια εξέλιξη, ελπίζω να μην ε, τα παραφουσκώσει ο τύπος. Γιατί Καλό θα είναι να μην έχει ο Βρετανό ε, υπήκο την εντύπωση ότι εκεί που κάθεται στο λεωφορείο θα έρθει να του χτυπήσει την πλάτη ένα ε, για να τον καλέσει στι Βρυξέλλε στην Και για να απαντήσω και στον κύριο Μπρόντ, συμφωνούμε ότι δεν υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προσέλευση, δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιβάλλει κυρώσεις, οι εθνικές αρχές μέσω των εθνικών αρχών θα μπορέσουμε να ε, επιβάλλουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, στην περίπτωση της Βρετανίας, εάν ένας Βρετανός υπήκος αρνηθεί κατά τρόπο να δικαιολόγητο κατά την άποψή μας να ε, προσέλθει, θα ζητήσουμε από τις αρχές της Βρετανίας να εξετάσουν την υπόθεση αυτή. Δηλαδή ένα δικαστήριο καταρχάς θα κοιτάξει εάν ήταν δικαιολογημένη ή μη η άρνηση ε, μαρτυρίας ή προσέλευσης και στη συνέχεια εάν υπάρχει λόγος επιβολής Ρώσων. Δεν πρόκειται να επιβληθεί ένα υπερεθνικό ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο θα υπερκαλύπτει τα εθνικά στην περίπτωση αυτή. Για τον κύριο Ντάφ. Δεν έχω μιλήσει απευθείας με τον Ombudsman για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία από τη διαδικασία της Επιτροπής, αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, που στηρίζονται και απορρέουν από τους κανόνες που ισχύουν για το θεσμό του διαμεσολαβητή. Έχουμε εμπνευστεί λίγο πολύ από αυτό το θεσμό. Και με αυτήν την νέα εξέλιξη των διατάξεων και των διαδικασιών, εγώ δεν ε, διαγνώσκω ακριβώς σύγκρουση μεταξύ της Εξεταστικής Επιτροπής και του ε, διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι έχει ο καθένας διαφορετικές αρμοδιότητες και εξουσίες. Για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το άρθρο 475, τη σχετική ερμηνεία, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη σημασία εν προκειμένου. Ε, δεν έχει μεγάλη σημασία το πώς θα δοθεί ο όρκος αρκεί να δίνεται και να αντιλαμβάνεται ο πολίτης τη σημασία του. Ο τύπος ο συγκεκριμένος δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και μη λησμονούμε ότι μπορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να υπάρχει, αλλά υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που δεν γνωρίζουν αυτή την παράδοση στην νομική τους, αυτόν τον τύπο, δηλαδή τον, τον όρκο, την έναρξη μαρκετρία στην ε, νομική τους παράδοση. Όπως είπα, οι κυρώσει θα περνούν μέσα από, τον, ε, από τη διοικητική διαδικασία ενός κράτου μέλους και όπως και να έχει χρειάζεται διοργανική συμφωνία για να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα αυτό. Άρα θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν. Για τη δική σας ερώτηση, Πρόεδρε, που ήταν πολύ σημαντική επίσης. Ε, το ενδεχόμενο δηλαδή να ξεκινήσει μια δικαστική μια διαδικασία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια λειτουργία μια εξεταστική επιτροπή. Ε, εμείς έχουμε προβλέψει εδώ ότι μπορεί να αποφασίσει το Κοινοβούλιο να άρει τη λειτουργία, να διακόψει τη λειτουργία αυτή τη εξεταστική επιτροπή, όσο εκκρεμεί η υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων, ανάλογα βέβαια και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ε, υπόθεση ε, έχω προβλέψει λέει, δηλαδή, τη σχετική διάταξη στο κείμενό μου. Επίσης η Γραμματεία έχει εξετάσει την κατάσταση που ισχύει στα κράτη-μέλη και την έχουμε παρακολουθήσει λίγο πολύ. Θα ήθελα να δώσω κάποια παραδείγματα. Στο Βέλγιο Φερρυπίν ε, άρνηση μαρτυρίας μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση από 8 ημέρες σε 6 μήνες. Η ψευδορκία μπορεί ενώπιον εξεταστική επιτροπή μπορεί να οδηγεί σε φυλάκιση από τρει μήνε έω δύο χρόνια. Στη Γαλλία η άρνηση προσέλευση σε εξεταστική επιτροπή μαρτυρία μπορεί να οδηγεί σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή 7.500 ευρώ. Στο Λουξεμβούργο η ψευδορκία ή η δωροδοκία μάρτυρα μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση από δύο μήνες έως τριών ετών. Και αν διαβάζω σωστά, 123 3 ευρώ πρόσθεση μέχρι, μέχρι 7.436 ευρώ. Δεν ξέρω αυτή η ακρίβεια τι σημαίνει, αλλά έτσι μου λένε τα χαρτιά μου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ε, μελετήσει συγκριτικά την υπόθεση, αλλά εάν θέλετε να επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο την ε, γραμματεία, ώστε να έχουμε μια ε, εκτενέστατη εικόνα του τι συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη, δεν έχω αντίρρηση για το χρονοδιάγραμμα. Από τι άτυπε επαφέ μα, χωρίς όμω να μπορώ να πω τίποτε περισσότερο ε, προ το παρόν, ε, η Προεδρία τη Δανία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να προωθήσει το θέμα αυτό. Το πράγμα το οποίο μα βολεύει και ω προ το δικό μα χρονοδιάγραμμα, το ιστορικό. Δηλαδή, θα έχουμε περισσότερο περιθώριο για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και άρα, ίσω μπορούμε να φτάσουμε στην Ολομέλεια μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο για να περάσει στην προσεχή ε, προεδρία. Στη μεταπροσοχή Προεδρία συγκεκριμένα. Αλλά αυτά χονδρικά μόνο μπορώ να σας τα δώσω ως διάγραμμα. Και επίσης από τις άτυπες επαφές που είχαμε με την Επιτροπή και ευχαριστώ ιδιαίτερος τον Επίτροπο Σελκοβιτς για, την, ε, για, το ενδιαφέρον που έχει δείξει την υπόθεση αυτή. Και ιδιαίτερα, όπως είπα και από την αρχή, τη γραμματεία της Επιτροπής μας, γιατί εδώ και 4-5 μήνες ήρθα σε επαφή μαζί τους και στη συνέχεια όταν άρχισα να ε, σχεδιάζω την έκθεση συνεργάστηκαν μαζί μου και μου προσέφεραν το υλικό ακριβώς που χρειαζόμουν για να το ενσωματώσω στο κείμενο. Και έτσι έχουμε ένα κείμενο το οποίο τουλάχιστον αντιστοιχεί στους δικούς μου, στις μου προθέσεις και στόχους και ελπίζω στο τέλος και στις ε, προθέσεις και τους στόχους Μου φαίνεται λοιπόν ότι και εμείς με τη σειρά μας θα πρέπει να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα ο στόχος του εισηγητή είναι να προχωρήσει στη διατύπωση της ε, έκθεσής του σχετικά σύντομα και γι' αυτό μπορούμε να ορίσουμε κύριε Μάρτιν την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας την 11η Οκτωβρίου Οπότε στις 11 Ιουλίου η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών τα μεσάνυχτα της 14 Σεπτεμβρίου, πρώτη συζήτηση στις 19 Σεπτεμβρίου, δεύτερη συζήτηση στις 4 Οκτωβρίου και ψηφοφορία στις 11 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ευηθετικά, οπότε ε, ελήφθη πλέον η απόφαση, τελειώσαμε με το σημείο 7. και φτάνουμε στις ψηφοφορίες νομίζω. Δεν είναι ακόμα 10, αλλά φτάσαμε στις ψηφοφορίες. Ο κύριο Ταρκόφσκι, φτάσαμε στι ψηφοφορίε ή θα φτάσουμε στι ψηφοφορίε στι 10. Έχουμε 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Θα θέλατε να ξεκινήσετε εσεί και να διακόψουμε μετά τη συζήτηση. Καλώς λοιπόν. Τότε θα περάσουμε απευθείας στο σημείο 11. 15 συγγνώμη. Στο σημείο 15 Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο κ. Στακόφσκι θα μας παρουσιάσει το θέμα αλλά συμφωνούμε ότι όταν φτάσει η ώρα των ψηφοφοριών θα διακόψουμε. Κύριε Ταρακόφσκι, έχετε το λόγο. πρέπει να δώσουμε μια γνωμοδότηση για το ευρωπαϊκό εξάμεινο σε σχέση με την έκθεση ΕΚΟΝ, ε, η οποία έχει προετοιμαστεί από την Περβάνς ε, Περές και αφορά τον ε, συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών και την δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έγινε μια συζήτηση για το άρθρο 1 ε, για το άρθρο 121 και το άρθρο 136 που αφορά την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της, ε, των χωρών όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις γραμμές του προπολογισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη βάση της συνθήκης πρόκειται για τις χώρες μέλη που θα προετοιμάσουν τα εθνικά προγράμματα σύγκλησης, τα οποία θα αναθεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς το πρόβλημα ήταν ότι σε αυτή τη νέα άσκηση, η οποία ονομάζεται Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν δεν ε, λαμβάνεται παρκώς υπόψη με ένα ξεκαθαρό τρόπο. Και η Επιτροπή ΕΚΟΝ αυτό το οποίο κάνει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη ρύθμιση για, τον, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι να περιγράφει μια ρύθμιση για τις ε, διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε να καθοριστεί αυτή η διαδικασία και να ξεκαθαρίσει ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να υπενθυμίσω του συναδέλφου ότι ασχολούνται με μια τακτική διαδικασία του κανονισμού και τώρα ολοκληρώνουμε την πρώτη ανάγνωση στην ΕΚΟΝ. Ε, ήταν, ε, χθες έγινε η πρώτη τριμερή συνάντηση. Η βασική ιδέα είναι να συμπεριληφθούμε στη διαδικασία όλες, σε, και στις τρεις φάσεις. Καταρχήν, να υπάρξει μια μεικτή διακοινοβουλευτική επιτροπή όπου θα υπάρξουν μέλη τη Επιτροπή Απασχόληση, Προπολογισμού και τη ΕΚΟΝ και να αναλάβουν σημαντικό ρόλο και στι τρει φάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτή, αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα γίνεται κάθε χρόνο, θα υπάρξει μια φάση συντονισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ότι πρώτα ο Επίτροπο, ο οποίο είναι υπεύθυνο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα θέτει ερωτήσει προ την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Μια άλλη πρόταση είναι να συσταθεί μια διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών εθνικών, των Εθνικών Κοινοβουλίων και θα έχουμε ένα ψήφισμα για την στρατηγική Ευρώπη 2020 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα απαντήσει κάποιες ερωτήσεις από το σώμα. Αυτό θα είναι ο ρόλος μας στη φάση του συντονισμού. Στη συνέχεια υπάρχει η φάση παρακολούθησης όπου θα οργανώσουμε σχεσμένα εργαστήρια, workshops, ακροάσεις όπου οι χώρες ε, μέλη βρίσκονται στη διαδικασία να οριστικοποιήσουν τα προγράμματα σταθερότητας και ε, σύγκλησης και θα τα συζητήσουμε. Η ΕΚΟΝ θα οργανώσει πάνελ με πυρογνώμονες για την οικονομική εποπτεία και η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες ε, γραμμές της, Επιτροπή, θα τις δημοσιοποιήσει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και στο Κοινοβούλιο. Και στη συνέχεια θα υπάρξει μια τρίτη φάση. Ε, και μετά από συζητήσεις με τους συναδέλφους που πραγματεύτηκαν όλα αυτά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δύο αυτές ε, φάσεις ε, μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Υπάρχουν ξεκάθαρα αιτήματα από τη δική μας πλευρά, τα οποία έγιναν δεκτά και από τα τρία θεσμικά όργανα. Το πιο επίμαχο θέμα και το πιο σημαντικό σχετίζεται με την τρίτη φάση της πρότασης που αφορά τη λεγόμενη παρακολούθηση, το follow-up. Και εμείς προτείνουμε κάτι το οποίο μια, ε, είναι σαν άσκηση λογοδοσίας, όπου οι χώρες μέλη καλούνται να εξηγήσουν τις πολιτικές του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα οργανώσουμε και μια συζήτηση με επικεφαλής των κυβερνήσεων πριν από την ε, οριστικοποίηση των μηχανισμών σταθερότητας. Οι διάφορες ε, χώρες ε, μέλη θα παρουσιαστούν λοιπόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επικεφαλείς και θα εξηγήσουν την, τις πολιτικές τους. αν υπάρχει μια κινητοποίηση μηχανισμών σταθερότητας, το Συμβούλιο θα πρέπει να δικαιολογήσει τη δική του θέση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό είναι το πιο επίμαχο θέμα, το μείζον θέμα το οποίο συζητείται εντό αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι είναι το πιο, η πιο σκληρή απόφαση η οποία να ληφθεί. Το άλλο σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί και μα αφορά ε, ω Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων είναι με ποιο τρόπο θα πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η σχέση γιατί το Συμβούλιο και κατά κάποιο τρόπο η Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, θέλουν να το κάνουν μέσω του κανονισμού. Ενώ το δικό μας αίτημα είναι να υπάρχει μια διοργανική συμφωνία εν σχέση με το θέμα αυτό και σε σχέση με την ρύθμιση αυτή τη σχέση, τη μόρφωση της σχέσης. Ε, και η ε, ο τερμερής διάλογος ε, έγινε χθε όπως σας είπα και πάμε προς ένα συμβιβασμό γιατί τα περισσότερα από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για μας συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό αλλά υπάρχουν πολιτικές εμάδες που εμένουν, εξακολουθούν να εμένουν στη διοργανική συμφωνία. Ανακύπτει ένα θέμα για τη δική μας γνωμοδότηση, κατά πόσο θέλουμε να συμπεριληφθεί εδώ και τι θα πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί η θέση του Κοινοβουλίου, όπως δηλώνεται από την ΕΚΟΝ, που είναι η αρμόδια επιτροπή, έχει διατυπωθεί. Αλλά υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις σε σχέση με έναν ήπιο μηχανισμό συντονισμού για το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πιο πλατιά συζήτηση για το ρόλο αυτών των εργαλείων σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Επίσης για την Νομική Επιτροπή η οποία εξάδεσε μια γνωμοδότηση αλλά είναι και ένα θέμα νομικής βάσης. Ε, ξέρετε ότι υπάρχει θέση ότι θα πρέπει να επιλέξουμε μία βάση ε, της συνθήκης. Και υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δύο βάσεις της συνθήκης ταυτόχρονα το 1.21 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί το 1.36 λέγεται από την Νομική Επιτροπή. Και νομίζω ότι υπάρχει εν γέννη ένα συνταγματικό θέμα σχέση με αυτά τα θεσμικό όργανα. Δεύτερον, για τη θέση του Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο, ε, κατά πάσα θα πρέπει να ενισχυθεί και τρίτον ε, το θέμα της βάσης της συνθήκης και πώς θα πρέπει να επιλεγεί, αν είναι μία ή δύο. Ε, αυτά είναι τα θέματα τα οποία μένουν ανοιχτά προς συζήτηση και είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε τάχιστα τη συζήτηση γιατί όπως σας είπα περιμένουμε η πρώτη ανάγνωση σύντομα να ολοκληρωθεί. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Α, συγγνώμη, δεν διάβασα καλά. Πρώτα έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό εμείς να εκφέρουμε μια γνωμοδότηση, να συντάξουμε μια γνωμοδότηση καλύτερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όπως είπε ο κ. Στακόφσκι, πέρα από το σημαντικό θέμα του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που έχει ήδη τεθεί στα πλαίσια της έκθεσης Μπερές, νομίζω ότι το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ανακοινεί και θέματα, θα έλεγα, γενικότερα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει ένα περίεργο, θα έλεγα, νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο τεχνικά δεν ρυθμίζεται από μία ή αδίποτε ρύθμιση ενός ας πούμε κώδικα συμπεριφοράς ε, που ορίζεται στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας. Αντίθετα, στα πλαίσια των δύο ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατέθεσαν την πρόταση, θεωρείται το σημείο αυτό σαν ένα σημείο σύνθεσης και συντονισμού των διαφόρων πλευρών της οικονομικής διακυβέρνησης και του, ε, δημοσιονομικού και της μακροοικονομικής σταθερότητας και της στήριξης στην ανάπτυξη. Τρεις, πιλότες, ε, τρεις ε, συγγνώμη, πυλώνες που βρίσκονται κάτω από την στρατηγική 2020. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια σύνθεση του συνόλου των μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση και η διαχείριση του εξαμήνου επαφίεται σε ένα κώδικα συμπεριφοράς που προβλέπεται για έναν από τους πυλώνες αυτούς, δηλαδή το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ενώ είναι προφανές από τις συνθήκες ότι τα κράτη-μέλη συντονίζουν τις οικονομικές τους πολιτικές στο εσωτερικό της Ένωσης, όπως λέει το άρθρο 5, και όπως λέει το άρθρο 121.6 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ρυθμίζουν τις διάφορες μορφές εποπτείας και διακυβέρνησης μέσα από συγκεκριμένους κανονισμούς. Θα πρέπει η Επιτροπή μας λοιπόν να αντιμετωπίσει το θέμα του θεσμικού ε, καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να προσδώσει εν πάση περιπτώσει ένα τέτοιο καθεστώς νομικά καθορισμένο και να πω ότι ενώ στην έκθεση Μπερές λέγεται ότι το εξάμεινο θα πρέπει να ρυθμίζεται από ένα κανονισμό ή από μια διαθεσμική συμφωνία Τώρα στα πλαίσια αυτής της πρώτης ανταλλαγής απόψεων εμείς θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με το 126.6 απαιτείται να υπάρξει ένας κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Παράλληλα πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδεσμεύσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο από την άμεση σχέση με μία από τις πλευρές της διακυβέρνησης, δηλαδή το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αν το κάνουμε αυτό τότε θα μπορέσουμε να διορθώσουμε και έναν στόχο ο οποίος θα διασφαλίσει την ισορροπία του προτύπου το οποίο επιδιώκουμε. Από τη μία λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει και λιτότητα και από την άλλη ανάπτυξη, αλλά παρόλα αυτά ε, διευκρινίζουμε τα μέσα για να το πετύχουμε μόνο ως προς τη λιτότητα και όχι ως προς το δεύτερο που είναι η ανάπτυξη. Συνεπώς θα πρέπει λοιπόν εμείς να αποδεσμεύσουμε το εξάμεινο από μία εικόνα ε, που δίνει ότι στην ουσία είναι παιδί του Συμφώνου Σταθερότητας και θα πρέπει να το συνδέσουμε με το σύνολο των οριζόντιων πολιτικών της Ένωσης όχι μόνο στα πλαίσια της νομικής του βάσης αλλά και στα πλαίσια της πολιτικής του αξίας δηλαδή να αξιοποιήσουμε την ιδέα ότι η οικονομική πολιτική της Ένωσης είναι ένα σύνολο πολιτικών που συνοντίζονται και μεταξύ τους σε επίπεδο οριζόντιο πολιτικές σταθερότητας από τη μία, αναπτυξιακές πολιτικές από την άλλη είτε σε κάθε το επίπεδο από τη μία οι πολιτικές των κρατών μελών και από την άλλη οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ τίθεται και το θέμα του προϋπολογισμού της Ένωσης και των διαφορετικών πολιτικών που πρέπει να γίνονται αντικείμενο συντονισμού με τις πολιτικές των κρατών μελών. Η πολιτική της Ένωσης δηλαδή συντίθεται από τις πολιτικές των κρατών μελών και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός αυτών των κάθετων και οριζόντιων πολιτικών είναι η κοινοτική Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και γι' αυτό πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αυξήσει το ρόλο του, θα πρέπει το εξάμεινο αυτό να είναι εξάμεινο των κοινοβουλίων και όχι μόνο κυβερνήσεων και να ελέγξουμε σωστά τον τρόπο λειτουργίας του κανονισμού του εξαμήνου. Έχουν ζητήσει το λόγο ο κύριος Νταφ και ο κύριος Μπρόνς. Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει στην ώρα των ψηφοφοριών. Αλλά εάν ο κύριος Μπρόντς και ο κύριος Ντάφ μπορέσουν να μιλήσουν σχετικά σύντομα, τότε ίσως να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό τώρα, καθυστερώντας λίγο την αρχή των ψηφοφοριών. Λοιπόν, τότε θα διακόψουμε, όχι ο κύριος Ντάφ θα ήθελε περισσότερο χρόνο, οπότε ε, θα διακόψουμε, θα συνεχίσουμε μετά τις ψηφοφορίες με τους Νταφ και Μπρόντς. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες.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 Γι' αυτό ξεκινάμε. Θέτω καταρχάς σε ψηφοφορία την τροπολογία 12. Α, όχι. Τη συμβιβαστική τροπολογία Α. Ο κύριος Νταφ. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, να πω δύο λόγια πριν αρχίσουμε τη ψηφοφορία. Πολύ σύντομα. Και θα ήθελα να ευχαριστώ καταρχά του συναδέλφου από τι άλλε ομάδε για το πνεύμα συνεργασία μέσα στο οποίο καταλήξαμε σε αυτέ τι συμβαστικέ τροπολογίε. Πολύ συγκεκριμένα, στην υπαριθμόν C γάμα, συμβαστική τροπολογία, ο κ. Φωτοκρής έχει μια προφορική τροπολογία. Στη σελίδα 3 μπορείτε να τη διαβάσετε. και ζητεί την ενσωμάτωση της διάταξης ότι μπορεί μια πολιτική ομάδα να ζητήσει σύγκληση εξεταστικής επιτροπής. Ε, σύγκληση της επιτροπής, συγγνώμη. για την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης. Όπως εγώ έχω συντάξει το κείμενο, την ε, σύνταξη αυτής της αξιολόγησης ε, την αναλαμβάνουν οι συντονιστές και η Επιτροπή στην ολομέλειά της ε, συνέρχεται μόνο σε περίπτωση που δεν μπορούν να καταλήξουν συμφωνίες συντονιστές. Όμως ο συντονιστής εκπροσωπών πολιτική ομάδα και συντονίζουν εκ μέρου πολιτικής του ομάδας νομίζω ότι ούτως ή άλλως αυτή τη δουλειά έχει να κάνει και έτσι το να συμπεριλάβουμε το συγκεκριμένο αυτό αίτημα ε, για πρωτοβουλία πολιτικής ομάδας είναι και πλεονασμός. Πέραν αυτού, όμως, ανοίγει και το, την προοπτική Αρχέ μη νομιμοποιούμενες, δηλαδή γενικοί γραμματεί των πολιτικών ομάδων που δεν έχουν ρόλο στην διαδικασία ακρόασης και επικύρωσης της υποψηφιότητα ενός επιτρόπου, να παρεμβαίνουν πολιτικά την τελευταία στιγμή. προκειμένου να ελέγξουν έναν υποψήφιο επίτροπο. Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, αλλά και πιο διεξοδική και προσεκτική στη δουλειά της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθεί η διαδικασία έγκρισης. Έτσι λοιπόν θα πω στον ε, κύριο συνάδελφο ότι δεν πρόκειται να αντιταχθώ στην ε, υποβολή της προφορικής τροπολογίας προς ψηφοφορία, γιατί σέβομαι το δικαίωμά του να καταθέτει προφορική τροπολογία, αλλά εγώ προσωπικώς και η ομάδα μου των φιλελευθέρων θα καταψηφίσουμε την τροπολογία αυτή. Ο κύριος Φόξ ζητεί μια ε, χωριστή ψηφοφορία για τη δέσμευση δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρους τους οποίους ζητεί να διαγραφούν από το κείμενο. Εγώ όμως θα επιτρέψω την προφορική τροπολογία μεν, αλλά ε, θα καταψηφίσω την πρόταση, διότι δεν μπορεί όροι που βρίσκονται στη συνθήκη, δεσμεύσει δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαγραφούν. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων προς εσάς κύριε να που θα σε αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Θα, θα, θα προσπαθήσω να αντιταχθώ στις υπόνοιε υπόνοιές σας. Η έννοια της τροπολογίας ε, έχει ως εξής έχουμε πάντοτε τη δέσμευση να συγκαλούνται οι συνεδριάσεις της Επιτραπής. Μετά από αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες, γιατί δεν πρόκειται για την πρακτική, στην ουσία δίδεται μεγαλύτερη εξουσία στους συντονιστές. αλλά η έκβαση μπορεί να είναι διαφορετική. Σε μια περίπτωση μπορεί η απόφαση να είναι εύκολη και είναι σωστό να μην συγκαλείται η συνεδρίαση της Επιτροπής. Από την άλλη μπορεί να πρόκειται για μια σκληρή απόφαση και στην περίπτωση αυτή μπορεί να συγκληθεί η Επιτροπή. Αλλά είναι σκληρή η απόφαση όταν υπάρχει συμφωνία προς την απόφαση αυτή αλλά θέλουν να, επιθυμούν να συγκληθεί η συνεδρία της Επιτροπής για να επικυρώσει αυτή την απόφαση. Και αυτό είναι απολύτως θεμητό. Είναι θεμητό να, οι πολιτικέ ομάδες να παρέμβουν για να συγκληθεί μια συνεδρίαση της Επιτροπής ούτω ώστε να επικυρωθεί μια δύσκολη απόφαση. Ε, φυσικά πάντοτε γίνονται πολιτικές διαβουλεύσεις και δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Ε, θεωρώ ότι οι τροπολογίες πραγματικά ε, παρέχουν πλατιές δημοκρατικές δυνατότητες για αυτού του είδους διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θέτω σε ψηφοφορία την συμβιβαστική τροπολογία α. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές καταπίπτουν συνεπώς οι τροπολογίες 12 και 1. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ένα είναι κατά. Δεκτή. Τροπολογία 14. Γουερέρο Σαλόμ. Ποιοι είναι υπέρ. κατά. Απορρίπτεται. Το προ... Τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή ομόφωνα. Φτάνουμε τώρα στην τροπολογία 15. Όχι, έχουμε φτάσει στην τέταρτη συμβιβαστική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές ομόφωνα δεκτή, οπότε καταπίπτουν οι επόμενες τοπολογίες και φτάνουμε τώρα στη συμβιβαστική Β. όχι, για μια στιγμή. Όχι, ναι, συμβιβαστική Β επανέρχεται ο πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ. Α, Συγγνώμη, συγγνώμη, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει ο πρόεδρος. Για μια στιγμή. Έχει ζητηθεί από τον κύριο Φόξ να υπάρξει και χωρισμένη ψηφοφορία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση μέχρι εκεί. Ποιοι είναι υπέρ του να μείνει αυτή η μικρή φράση. Ποιοι είναι κατά της ευρωπαϊκής υποχρέωσης. Γίνεται δεκτή. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για το υπόλοιπο κομμάτι της τροπολογίας. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτή. Πηγαίνουμε στο 17 τώρα. Μέσερ Σμιτ ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν απορρίπτεται. Οι 18 ποιοι είναι υπέρ. κατά δεκτή 10 υπέρ 9 κατά φτάνουμε τώρα στην τροπολογία 10 α, έχει καταπέσει 7 μάλλον έχει αποσυρθεί 8 φτάνουμε στην 19 ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ κατά αποχές δεκτή. Τώρα φτάνουμε στην βιβαστική ε, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Καταπίπτυρη 9. Φτάνουμε στην τρίτη συμβιβαστική. Έχει ζητηθεί και εδώ και χωρισμένη ψηφοφορία. Όχι, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει όμως μια προφορική τροπολογία Σαουντάργα, στην οποία θα ψηφίσουμε πρώτα. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας Σαουντάργας. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα το δεύτερο τμήμα, το σύνολο ουσιαστικά του κειμένου. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δεκτή. Οι επόμενες τροπολογίες έχουν όλες καταπέσει. Και πάμε απευθείας στην τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Φτάνουμε στην τελική ψήφο. Ποιοι είναι υπέρ. κατά 18 υπέρ 1 κατά δεκτή. Συγχαρητήρια για την ευτυχή κατάληξη της προσπάθειας την οποία έκανε ο συνάδελφος Άντριο Νταφ. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για την καλύτερη νομοθετική δραστηριότητα, επικουρικότητα, αναλογικότητα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τον συνάδελφο Μέσερ Σμιτ να μας παρουσιάσει τις θέσεις του για τις τροπολογίες πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τη Γραμματεία για τη βοήθειά τους. Νομίζω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια διατύπωση έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι όλες οι τροπολογίες μπορώ να αντισυστήσω συστήσω έγκριση ευχαριστώ Λοιπόν, μιας και ο εισηγητής είναι υπέρ όλων των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί, κυρίως από τον συνάδελφο Ράντζελ και από τον συνάδελφο Σόλτς, Μορέιρα, Νταφ, Γέτερμακη και τα λοιπά. Όλες εν πάση περιπτώσει τις τροπολογίες τις δέχεται ο εισηγητής και μπορούμε να τις ψηφίσουμε ομαδών, ο κύριος Νταφ. θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια τέτοια ψηφοφορία, να κάνουμε μια τέτοια ψηφοφορία, αλλά η τροπολογία 10 του κυρίου Μορέιρα λέγει και ίσως να είναι γλωσσικό βέβαια το θέμα και όχι θέμα ουσίας. Λέγει όμως ο κύριος Μορέιρα στα αγγλικά τουλάχιστον ότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιπτώσεων είναι κάτι το υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, αλλά δεν είναι, λέει ο κύριος Νταφ. Είναι κάτι το επιθυμητό, το ευκταίο, αλλά υποχρεωτικό δεν είναι. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να προτείνω να πούμε ότι ε, είναι όχι υποχρεωτικό, δεν είναι σωστό, αλλά επιθυμητή. Στο δικό μου κείμενο, λέει ο κύριος Μέσερσμιτ, το νόημα είναι ότι είναι κάτι το επιθυμητό. Ο κύριος Νταφ λέει ότι δεν, ε, δεν ομιλώ την γλώσσα της Δανίας, λέει ο κύριος Νταφ. Και ο κύριος Μπρόκ λέει ότι η γλώσσα της Δανίας δεν είναι γλώσσα. Λοιπόν, θα δούμε. Μιας και υπάρχουν από ό,τι φαίνεται προβλήματα Ας ψηφίσουμε λοιπόν ο μπλοκ τις πρώτες τροπολογίες και μετά θα ψηφίσουμε ε, ε ομαδών όλες τις τροπολογίες μέχρι την 10 όπου τέθηκε το θέμα και μετά τις δύο τελευταίες. Λοιπόν ψηφίζουμε πρώτα την 1, 2 και 3. Ποιοι είναι υπέρ της 1, 2 και 3. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Τώρα 13, 14 και 15. Ο κύριος Ταρκόφσκι έχει ζητήσει μια... Έχετε κάποιο πρόβλημα ή θα τις θέσω σε ψηφοφορία και τις τρεις μαζί. Α, μία προς μία. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία τότε την τροπολογία 13. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος, για την 13. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Δεκτή. 10 υπέρ, 8 κατά. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Η ίδια κατάσταση δεκτή και η 14. 15. Ποιοι είναι υπέρ. Ομόφωνα δεκτή 15. Ο κύριος Ντάφ θέλει το λόγο. Όχι. Α, δεν υπήρχε ομοφωνία για την 15, μία διευκρίνηση λέει ο κύριος Ντάφ. Νομίζω ότι με δημοκρατικό τρόπο εξέφρασα τη διαφωνία μου, λέει ο κύριος Ντάφ. Λοιπόν, δεν έγινε δεκτή η 15 ε, ομόφωνα, αλλά με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία των τροπολογιών 4, 5, 6, 8, 9, ως εκεί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, δεκτές, για την 10 θα ήθελα να καταλάβω λίγο το θέμα που έθεσε ο κύριος Νταφ. Θα ψηφίσουμε απευθείας. Τι ακριβώς θέλετε κύριε Νταφ. Ο κύριος Μορέιρα λέγει ότι εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ε, έρευνας ε, συνεπειών είναι κάτι το υποχρεωτικό. Δεν είναι έτσι όμως. Η συνθήκη δεν το λέγει αυτό. Αντίθετα η συνθήκη λέγει ότι είναι μια επιθυμητή πρακτική την οποία σε αυτή τουλάχιστον την φάση το Κοινοβούλιο δεν τηρεί επίσημα. Προτείνω λοιπόν αντί να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη υποχρεωτικό, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ευκταίο. Θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή ότι το πρόβλημα το οποίο περιγράφει ο Άντριο Ντάφα στη γερμανική διατύπωση κατά την άποψή μου δεν υφίσταται γιατί η φράση εκφράζει λέει τα εξής Συγγνώμη, λέει ο μιλητή, έχασα τη σειρά, τη γραμμή. Εκφράζεται η επιθυμία να περιγράφεται αυτό δεσμευτικά. Αλλά δεν λέγεται ότι είναι δεσμευτικό. Εκφράζεται η επιθυμία να είναι δεσμευτικό. Sì, sembra che vi sia testo originale E dice obbligatoria? Eh? Sì, è obbligatoria, quindi la propositività è pertinente. Quella commissione d'accordo. Sì, commissione d'accordo. Allora, eh, il testo originale... Λοιπόν, το αρχικό... Α, ο Messerschmitt έχει ζητήσει το λόγο. Δεν έχω καμία αντίρρηση με την ε, ρύθμιση που προτείνει ο κ. Ταφ. Μπορούμε να αλλάξουμε τη λέξη. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Μωρέρα, αλλά για μένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Από την άλλη, εμείς είμαστε οι αρμόδιοι, έτσι και αλλιώς το αρχικό κείμενο φέρεται η αγγλική γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα. Το θέμα δεν είναι λοιπόν μετάφρασης, αλλά γενικότερα γλωσσικής ρύθμισης. Λοιπόν, θα αντικαταστήσουμε τη λέξη υποχρεωτικό από τη λέξη ευκταίο. Πρόεδρε, ο κύριος Γκουαλτιέρη, διαβάζοντας, λέει ο κύριος την Ιταλική διατύπωση πράγματι λέγεται κάτι το διαφορετικό. Δεν αναφέρεται ούτε στον υποχρεωτικό χαρακτήρα, το mandatory στα αγγλικά, και είναι λάθος, αλλά ούτε και ευκταίο, λέει απαραίτητο στα Ιταλικά. Λέει ότι είναι κάτι το πολιτικά απαραίτητο και όχι νομικά απαραίτητο. Το να κάνουμε λοιπόν μια τέτοια μεταφορά νοήματος από το απαραίτητο σε υποχρεωτικό είναι κάτι το λανθασμένο. Μπορούμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο είναι ναι μεν πολιτικά απαραίτητο αλλά θεσμικά όχι δεσμευτικό, όχι υποχρεωτικό. Δεν ξέρω τώρα όλα αυτά τα λέμε ενώ ο Μορέιρα δεν είναι παρόν. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του αλλά εν πάση περιπτώσει Κοιτάξτε, αν λέτε απαραίτητο, απαραίτητο σημαίνει και ευκταίο έτσι κι αλλιώς. Παρακαλώ, συμφωνήσουμε κάποτε, εν πάση περιπτώσει. Ο Γκουαλτιέρη προτείνει την αντικατάσταση της λέξης υποχρεωτικό από το πολιτικά απαραίτητο. Ο Νταφ προτείνει τη χρήση του επιθέτου ευκταίου. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ ε, της πρότασης του Νταφ γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε να το κάνουμε ουσιαστικά υποχρεωτικό. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ μακριά η πρόταση Νταφ από την άποψη του κυρίου Γκουαλτιέρη. Πάντως η αγγλική λέξη mandatory δεν είναι η σωστή. Το indispensable στα αγγλικά βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά διφορούμενο. Είναι μια έξυπνη λέξη εδώ. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με το επίθετο indispensable, απαραίτητο στα αγγλικά. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, αλλά δεν αλλάζουμε την ουσία, εν πάση Σήμερα έτσι και αλλιώς η διαδικασία αυτή αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωτική. Bene, allora la proposta anche dal punto di vista linguistico si dice Λοιπόν, από γλωσσική άποψη η πρόταση είναι καλύτερη στην Ιταλική γλώσσα, η λέξη απαραίτητο δηλαδή. Ψηφίζουμε την τροπολογία 10 λοιπόν, τροποποιημένη. Είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεχτή. 12 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην τελική ψήφο. Την 11 την ψηφίσαμε μόλις τώρα και την 12... Α, για μια στιγμή. Λοιπόν, 11 και 12 ξαναψηφίζουμε μαζί. 11 και 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο του κειμένου. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτό συγχαρητήρια στο συνάδελφο Μέσερ Σμιτ. Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη σας έκθεση κύριε Μέσερ Σμιτ. Ο Μέσερ Σμιτ δεν ακούει. Λοιπόν τώρα, ε, τι θα, πού πάμε τώρα ρωτάει ο πρόεδρος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 μετά από τη συζήτηση που ξεκινήσαμε χθε, διατυπώσαμε μία επιστολή προς τον πρόεδρο Μπούζεκ για την εκλογή του αντιπροέδρου. Δεν θα περάσουμε στις λεπτομέρειες, αλλά στην τελική πρόταση, στην τελική διατύπωση της επιστολής, μπορώ να σας διαβάσω το σημαντικό κομμάτι λίγο πριν από το τέλος. Εάν ένας μόνο αντιπρόεδρος πρέπει να αντικατασταθεί και εφόσον δεν υπάρχει παρά μόνο ένας υποψήφιος, ο υποψήφιος αυτός μπορεί να εκλεγεί διαβοής. Ο πρόεδρος έχει την διακριτική αρμοδιότητα να αποφασίσει για την χρήση της διαβοής μεθόδου ή και της μυστικής ψηφοφορίας εφόσον αυτός το κρίνει χρήσιμο. για την κάλυψη ε, του αντιπροέδρου ο οποίος, του οποίου η θέση χειρεύει. Λοιπόν, συμφωνείτε ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή η πρόταση που κάνουμε στην επιστολή αυτή και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το 13 ερμηνεία των άρθρων 50 και 51 στην περίπτωση συμφωνιών Α, συγγνώμη, όχι, αυτό ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά στην επεξεργασία του και γι' αυτό έχει αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη και συνεπώς θα φτάσουμε τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με την έκθεση του κυρίου Ταρκόφσκη. Και μετά να περιμένουμε να έλθει η προσκεκλημένη μας. Έχουν ζητήσει το λόγο για την έκθεση Ταρκόφσκη ο κύριος Νταφ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Um, ναι, λέει ο κύριος Δάφ. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε έναν κανονισμό όσον αφορά το άρθρο 1.0.21.6. Νομίζω ότι αυτό απαιτεί από μας ε, η συνθήκη. Ε, αυτό λέει άλλωστε και η έκθεση. και οι πέντε προτάσεις του πακέτου της οικονομικής διακυβέρνησης. Το ερώτημά μου αφορά την ε, κατάσταση της συζήτησης στο πλαίσιο του διαλόγου. ο οποίος έγινε χθες το βράδυ. Προχωρά, θα φτάσουμε, θα καταλήξουμε τον Ιούλιο σε μια συμφωνία στο επίπεδο της πρώτης ανάγνωσης. Γιατί αν ισχύει αυτό θα πρέπει πριν από την Ολομέλεια θα πρέπει να έχουμε ένα κείμενο εκ μέρους της Επιτροπής. Και αν έχουν έτσι τα πράγματα, η ποιότητα του πακέτου θα βελτιωθεί. Βεβαίω, αν πάμε στη δεύτερη ανάγκη, θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα, ποια είναι η αίσθησή σα για το πού βρίσκονται τώρα τα πράγματα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι οδηγίε προ τα προς χώρε μέλη όσον αφορά τη μακροοικονομική πολιτική, τη μουσιονομική πολιτική κλπ. είναι προφανώ ε, συνεπάγονται μια απομάκρυνση από την ε, κυριαρχία των κρατών αυτών. Και νομίζω ότι έχουν εκχωρήσει ένα σημαντικό τμήμα της κυριαρχίας τους και του ελέγχου του προπολογισμού τους ε, οι χώρες μέλη. Ε, και ε, η δική μας ε, κυβέρνηση καθώς και η προηγούμενη και η παρούσα κυβέρνηση με σόφρονα τρόπο, συνήθως δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον κανονισμό για την κυβέρνησή μας, απέφυγαν την Ευρώπη στο τομέα αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερος παρεμβατικό όταν μας υπαγορεύσει κανείς ποια θα είναι η μακροοικονομική μας πολιτική, η φορολογική πολιτική κλπ. Προφανώ η διατύπωση που χρησιμοποιείται στην περίπτωση τη μεγάλη Βρετανία λόγω του opt-out είναι σύσταση και όχι οδηγία. Και στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν υπόκειται σε κυρώσεις εάν δεν ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις. Ωστόσο κατανοώ ότι θα υπάρξουν κάποιες προτάσεις ούτως ώστε να καλούνται οι υπουργοί της Μεγάλης Βρετανίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να λογοδοτούν για τυχόν αποκλήσεις από τις στάσεις αυτές. Η Βρετανική κυβέρνηση είπε μέχρι στιγμής ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει με αυτό, αλλά ενδεχομένω ε, θα ε, αναγκαστεί να το κάνει. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι θέσεις των άλλων χωρών που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ και που δεν έχουν τα, τη δυνατότητα του opt-out της Μεγάλης Βρετανίας και προφανώς έχουν μια υποχρέωση να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη εφόσον εκπληρώσουν τα κριτήρια. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι το λόγο λοιπόν, γι' αυτό ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Τακόσκι για να απαντήσει. Ωραία, Εάν ε, κατάλαβα καλά, και σε αυτό κάνει τα πράγματα τόσο δυσχερή, γιατί αυτό που προετοιμάζουμε είναι μια γνωμοδότηση για την έκθεση της Περβάνς Μπερές, όχι για τον κανονισμό. Αυτό σημαίνει, ε, και αυτό μπορεί να γίνει ε, όσον αφορά την έκθεση τη Περβάνη Μπερέ, μπορεί να γίνει ψηφοφορία του Σεπτέμβριου. Έχουμε χρόνο λοιπόν. Αλλά αν θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή στον εφαρμογή τον κανονισμό, ε, τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα. Προφανώς είτε η δική μας γνωμοδότηση θα πειράσει τον κανονισμό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά οι δικέ μου πληροφορίε από χθε, αλλά όχι σημερινέ πληροφορίε, είναι ότι πηγαίνουμε πρώτα προ μια συμφωνία ε, στο επίπεδο τη πρώτη ανάγνωση. Είμαστε πολύ κοντά στην επιτεύξη μια τέτοια συμφωνία. Αλλά βεβαίω δεν γνωρίζω την οριστική έκβαση αλλά νομίζω θα ολοκληρωθεί στην πρώτη ανάγνωση. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ψηφοφορία για την γνωμοδότηση αυτή, και πριν από το Στρασβούργο. Αλλά όπω είπα, ε, διαδικαστικά δεν ε, το κάνουμε αυτό. Δεν πρόκειται μια γνωμοδότηση για τον κανονισμό, αλλά για την έκθεση Περβάνου Μπερέ, όπου υπάρχει μια θέση του Κοινοβουλίου. Και προφανώ είναι δύσκολο και ακόμα πιο δύσκολο εάν ε, κινηθούμε προς την κατεύθυνση που πρότεινε ο κύριος Γκουαλτιέρη. Γιατί αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την λογική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα πράγματα θα γίνουν πιο δυσχερή. Γιατί μπορούμε να το προσπαθήσουμε. Αλλά οι αποφάσεις ελήφθησαν ήδη χθες και η δική μας προσπάθεια θα είναι περιττή. Να δούμε λοιπόν ε, κατά πόσο επετεύχθη συμφωνία ή όχι. Θα και να κρυφθούμε σε αυτή την ε, επιτροπή, γιατί έστω και αν έχει επιτευχθεί η συμφωνία, δεν έχει νόημα για μα κατά τη ουσία να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε όλο το θέμα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη ψηφοφορία τον Ιούλιο κιόλα. Ε, αλλά αν δεν έχει επιτευχθεί η συμφωνία, θα έπρεπε να επιταχύνουμε κάπως τα πράγματα και να κάνουμε κάποιες επίσημες ε, επαφές με τον εισηγή, ώστε να διατυπώσουμε επισήμως τη δική μας άποψη. Αλλά όπως είπα, ας, ας δούμε πρώτα τι έγινε ακριβώς και στη συνέχεια θα πάρουμε μια απόφαση σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Αλλά όπως σας είπα θα είναι αρκετά δύσκολο επισήμως να ασκήσουμε επιρροή σε όλη αυτή τη διαδικασία, ειδικά εάν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε έστω και αν η συμφωνία, έστω και αν ε, συμφωνούμε μάλλον, να αλλάξουμε την ε, λογική του εξαμήνου όπως πρότεινε ο κύριος Γκουαλτιέρη. Λοιπόν τώρα η διαδικασία ε, θα πρέπει να ορίσουμε λίγο το χρονισμό. Στην ουσία πρέπει να περιμένουμε κάποια γεγονότα που δεν εξαρτώνται από μας. Θα πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει με την Επιτροπή ΕΚΟΝ η οποία κανονικά θα πρέπει να αποφασίσει τον Σεπτέμβριο. Αν θέλουμε λοιπόν και εμείς να επηρεάσουμε θα έπρεπε να εκφέρουμε την άποψή μας τον Ιούλιο. Εφόσον λοιπόν συμφωνείτε μπορούμε να θέσουμε το θέμα αυτό στις 12 Ιουλίου αλλά αν μας προτείνει μια αλλαγή των ημερομηνιών ο εισηγητής τότε θα πρέπει να υπακούσουμε. Ο κ. Γουαλτιέρη έχει δει το λόγο. Δεν νομίζω ότι μια κάποια ρύθμιση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και σύνδεσή του δεν θα έχει νόημα στα πλαίσια μετά την έγκριση των έξι λεγόμενων προτάσεων. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι θέμα περιεχομένου, είναι θέμα μεθόδου. Εμείς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο, η αντίστροφη πλειοψηφία κτλ. Μια ολόκληρη σειρά μέτρων τα οποία πρέπει ακόμα να συζητηθούν. Λοιπόν, αν αυτός ο κώδικας συμπεριφοράς μετατραπεί σε κανονισμό, τότε δεν συμβαίνει τίποτα, δεν αλλάζει κάτι. Είναι λοιπόν δυνατό να πούμε ότι ο κανονισμός αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετά από την υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση του πακέτου διακυβέρνησης. Ναι, αλλά τότε τίθεται το θέμα πόσο μακριά θα πάμε όσον αφορά την γνωμοδότηση, γιατί η γνωμοδότηση έχει σε σκοπό να σχολιάσει την έκθεση της υπερβάσεω. Περέσε. μπορούμε να το κάνουμε βέβαια, αλλά πόσο μακριά θα πάμε αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είχαμε μία συζήτηση χθε με τον εισηγητή για άλλα θέματα, πάντα σε σχέση με τον κανονισμό που θα τα συζητήσουμε μια κάποια άλλη στιγμή αλλά μου είπε η κυρία Μπερέ στα πλαίσια των συζητήσεων που είχαμε ότι όσο την αφορά δεν έχει κανένα πρόβλημα να αναλάβει και για μετά το Σεπτέμβριο την απόφαση της δικής της Επιτροπής. Οπότε εμείς θα έχουμε τον χρόνο που απαιτείται για να υιοθετήσουμε την πρότασή μας στις 12 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω, μ' άκουσε ο εισηγητής. Με ακούσατε κύριε Ταρκόφσκι. Είπα ότι χθε συναντήθηκα με την κυρία Μπερές και μιλήσαμε και διάφορα άλλα θέματα και είπαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι την απόφασή σας αν θέλετε πάρτε τη και το Σεπτέμβριο γιατί με διατεθειμένη είπε η κυρία Μπερές να αναβάλω για λίγο καιρό. Λοιπόν το ξέχασα αυτό προηγουμένως να σας το πω γιατί αφορούσε η συνάντηση αυτή την τροποποίηση ενός άλλου άρθρου του κανονισμού που κάποια στιγμή θα κληθούμε να συζητήσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να αναβάλουμε λοιπόν τη συζήτηση του θέματος σας κύριε Ταρκόφσκι για τον μήνα σε επιτέμβριο. Συμφωνείτε? Bene, noi adesso avremmo ancora Λοιπόν, περιμένουμε. τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να θυμίσω ότι η επόμενη έκτακτη συνάντησή μας Λούλιο, θα γίνει στις 4 Ιουλίου, Τετάρτη Ιουλίου λοιπόν από τις 9.30 ε, θα ξεκινήσει η έκτακτη συνάντηση με την παρουσία της Πολωνικής Προεδρίας και η επόμενη τακτική μας συνάντηση προβλέπεται για τις 11 και 12 Ιουλίου. Και τώρα διακόπτουμε λίγο για να περιμένουμε την κυρία Γιώρικ, η οποία θα έρθει στις 11. Παρακαλώ μη φύγετε μακριά, διότι θα καθυστερήσουμε μετά. Θα μας παρουσιάσει τα επιτελεστέντα κατά την Ουγγρική Προεδρία. Η κυρία Γιώρεκ είχε έρθει και στην αρχή του εξαμήνου για να μας μιλήσει για το πρόγραμμά της. Τώρα θα κάνει τον απολογισμό, πρέπει να είμαστε παρόντες και να εκφράσουμε και τις δικές μας απόψεις. Λοιπόν, περιμένουμε 10 λεπτά την έλευση της κυρίας Γιώρικ. Allora riprendiamo la seduta e accogliamo con gioia la... Συνεχίζουμε καλωσορίζοντας την εκπρόσωπο της Ουγγρικής Προεδρίας, την κυρία Γιώρη. Όλοι γνωρίζετε την κυρία Γιώρη. Ήταν συναδελφός μας. Μετά ανέλαβε κυβερνητικές αρμοδιότητες στη χώρα της Είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε και στην Ουγγαρία και εδώ με την κυρία Γιώρη. Ήταν παρούσα και στην αρχή της Προεδρίας της και μας παρουσίασε τότε το πρόγραμμα, αυτό που ήταν το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Τώρα έρχεται κοντά στο τέλος της Προεδρίας για να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε αυτό το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θυμίζω ότι και μαζί με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, ασχοληθήκαμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα όπως την έκθεση Μπρόκου Αλτιέρη για την αναδιάρθρωση της συνθήκης, την αλλαγές σε συγκεκριμένα άρθρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας δώσω το λόγο και μετά ελπίζω να υπάρξει χρόνος για να τεθούν ερωτήσεις. Έχετε το λόγο κυρία Γιώργη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, λέει στα Ιταλικά η κυρία Γιώρη. Με πολύ μεγάλη χαρά α, ξαναήρθα στην Επιτροπή σας, αλλά θα συνεχίσω στη λίγουα φράγκα του 21ου αιώνα, την αγγλική γλώσσα. με κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά ξανά επιστρέφω στην Επιτροπή επίσης. Τον Ιανουάριο είμαστε μαζί με τον Υπουργό Μάρτινε ενώπιόν σας για την εκκίνηση της Ουγγρικής Προεδρίας και τώρα έρχομαι για να σας ενημερώσω για τα επιτεύγματα του εξαμένου μας. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια και παρατηρήσεις με βάση και τις δηλώσεις και τις κατευθύνες γραμμές του Υπουργού Μαρτσινή στην ακρόασή του εδώ. Και βέβαια είμαστε θέση σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Θα θυμάστε ίσως πως η Ουγγρική Προεδρία είχε επιλέξει ένα πολύ απλό σύνθημα, ισχυρή Ευρώπη. Και δεν λησμονήσαμε ποτέ και την διάσταση της σκληρής Ευρώπης με την ανθρώπινη πτυχή. Είμαι βεβαία ότι χάρη στις δραστηριότητες μας, ε, χάρη στις επιλογές μας, οι δραστηριότητες μας είχαν ως επικεντρό τον ανθρώπινο παράγοντα και ότι χάρη σε αυτές μπόρεσε να γίνει πιο ισχυρή η Ευρώπη. Επίσης, υποσχεθήκαμε και έτσι καθοδηγήσαμε και την Προεδρία μας, το εξέμεινο μας, να είμαστε μια Προεδρία με το βλέμμα στραμμένο προς το Κοινοβούλιο. Και είμαι βεβαία ότι και εσείς το διαπιστώσατε αυτό τους τελευταίους μήνες ότι η Προεδρία μας ήταν φιλικά προσκύμενη προς ε, το Κοινοβούλιο. Έγιναν πολλές διαβουλεύσεις και όχι μόνο υποχρεωτικές, όχι μόνο αυτές που είχαν να κάνουν με τα νομοθετικά, με την νομοπαραγωγική διαδικασία, αλλά και ε, διαβουλεύσεις που βελτίωσαν τις διοργανικές σχέσεις. Και είμαι βεβαίω ότι έχουμε και στο τομέα αυτό να επιτύχει σημαντική πρόοδο. Επίσης, και όχι μόνο λόγω της προσωπικής μου δέσμευσης ως πρώην Ευρωβουλευτού και πρέπει να σας πω ότι μερικές φορές είναι μεγάλη πρόκληση αλλά είναι και πολύ ωραίο να αλλάζει κανείς ε, ρόλο και να περνάει από την άλλη μεριά του τραπεζιού γιατί έτσι έχει μια ε, πιο συνολική εικόνα της κατάστασης. Ήταν επιλογή λοιπόν όχι δική μου μόνο και λόγω της προσωπική μου εμπειρία, αλλά και της κυβέρνησή μου, του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Η κυβέρνησή μας λειτουργήσε με βάση αυτήν την προοπτική και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη της απόψεις του Κοινοβουλίου. Γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου του Κοινοβουλίου καθώς και την, ε, τις εξελίξεις θεσμικές οι οποίες πλέον ισχύουν μετά τη θέση ενισχύ της ε, Συνθήκης Λισαβόνας. Άρα, μια ισχυρή Ευρώπη, σχέσεις καλές με το Κοινοβούλιο, δηλαδή καλύτερες διοργανικές σχέσεις για να επιτύχουμε το στόχο της χειρότερης Ευρώπης. Τι σημαίνει ισχυρή Ευρώπη. Η ισχυρή Ευρώπη σημαίνει γερονόμισμα, θεσμοί που συνεργάζονται και μεταξύ του και ισχυρε πολιτικές επιλογές χωρί να θέλω να επισέλθω στις λεπτομέρειες ενώπιον σας επί τη ουσία αυτών των επιλογών, επιλογών θα ήθελα να επισημάνω την ε, όθηση που δώσαμε σε μια συμφωνία για την οικονομική διακυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση του ευρώ, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενέργεια και την πολιτική συνοχή για την κοινή γεωργική πολιτική με στόχο να. Επειδή ε, μάλλον είμαστε πεπισμένοι ότι τέτοιες ισχυρές πολιτικές ενισχύουν την Ευρώπη, και η εσωτερική σχέση της Ευρώπης την καθιστά και πιο ανταγωνιστική στην ε, διεθνή σκηνή. Φυσικά δεν μπορώ τώρα να προβώ σε μια τελική αξιολόγηση. Μας μένουν ακόμη 15 μέρες. Μπορείτε να μου πείτε 15 μέρες δεν είναι τίποτα, αλλά δεν ισχύει αυτό στη δική μας περίπτωση. Αυτές οι 15 μέρες έχουν πολλά πράγματα. Έχουμε το, το six pack, το, την δέσμη των έξι μέτρων. Σήμερα το απόγευμα ξεκινάει με τον τριμερή διάλογο. Έχουμε επίσης ε, το θέμα των διαπραγματεύσεων για την Κροατία και την προσχώρησή της που το την Παρασκευή θα πρέπει να συστήσει στο Συμβούλιο στο τελευταίο σχέδιο κοινών θέσεων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα της προσχώρησης της Κροατίας. Άρα είναι πρόωρο ακόμη να ε, διατυπώσω συμπεράσματα και μια και δεν έχω ε, κρυστάλλινη μπάλα, δεν μπορώ να κρυστάλλινη σφαίρα, δεν μπορώ να προβλέψω τι θα προκύψει από αυτέ τι διαπραγματεύσει, αλλά θέλω να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την υποστήριξη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο ε, εξ αρχή για την προσχώρηση της ε, Κροατία. ήταν πάντα ένθερμο υποστήριξη στο Κοινοβούλιο και βεβαίω θα επισημάνω ότι και στο θέμα του ΣΥΚΣΠΑΚ ήμασταν πάντοτε σε συνεργασία με τους εισηγητές ε, για τα μέτρα αυτά και πάντα προσπαθήσαμε οι θέσει του Συμβουλίου να λαμβάνουν υπόψη και τις απόψεις του Κοινοβουλίου πριν να ε, διατυπωθούν τελικά και οριστικά. Μια τελευταία γενική παρατήρηση. Όλοι θυμόμαστε ότι η χρονιά ξεκίνησε με ένα αίσθημα δυσφορίας και απογοήτευση από πλευρά του Κοινοβουλίου. Εγώ ως πρώην Ευρωβουλευτής αντιλαμβανόμουν μάλιστα το λόγο αυτών των, αυτής της στις αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση για μια συνολική ανταπόκριση στην ε, κρίση ε, το Κοινοβούλιο αισθάνθηκε ότι είχε μείνει εκτός παιδιάς και ότι είχε αποκλειστεί από τη λήψη ζωτικών αποφάσεων. Η Προεδρία διαδραμάτισε ρόλο για την ενίσχυση της κοινοτικής μεθόδου και τώρα νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ πιο ξεκάθαρο και πιο υγιές πλέγμα διοργανικών σχέσεων. Και έτσι έχουν διασκεδαστεί οι αρχικοί φόβοι. Ξεκινώ με το θέμα της ε, μεταρρύθμισης συνθήκης, που ξέρω ότι απασχόλησε και τις συζητήσεις με τον ε, Υπουργό Μαρτινή τον Φεβρουάριο. Υπάρχει σαφή πρόοδο εδώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω ωστόσο ότι δεν ήταν διαδικασία που κίνησε η ίδια η Προεδρία. Αποτελούσε μόνο τμήμα αυτή τη συνολική ανταπόκριση στο θέμα της κρίσης το οποίο την κύρια ευθύνη φέρει το, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο, πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία, Πρόεδρε, να ευχαριστώ θερμά και και την ε, Επιτροπή σα για την πολύ ε, καλή συνεργασία. Γνωρίσαμε κάποιε δύσκολε στιγμέ το Μάρτιο και το Φεβρουάριο ήδη στην εξέλιξη αυτή τη υπόθεση. Ήμασταν σε διαρκή επαφή με του συγκητέ και μπορώ τώρα να σα πω με ιδιαίτερη ικανοποίηση πως Καταλήξαμε σε μια θετική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για το, με το ψήφισμά του. Καταλήξαμε σε μια θετική εξέλιξη στην μεταρρύθμιση αυτής επίπεδο Συμβουλίου και χάρη σε αυτές τις ε, κοινέ προσπάθειες, πιστεύω και της Προεδρίας μας αλλά και του Κοινοβουλίου, ε, μπορέσαμε να εισαγάγουμε ένα πολύ σημαντικό ε, κείμενο, μια πολύ σημαντική διάταξη στον Ευρωπαϊκό Σταθεροποιητικό Μηχανισμό προ το τρόπο λειτουργία του. Θα πρέπει δηλαδή το Κοινοβούλιο τακτικά να ενημερώνεται για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίηση. Το καταγράφω λοιπόν στα θετικά, στις επιτυχίες της κοινοτική μεθόδου. Ήταν μεγάλο επίτευγμα για μας. Το δεύτερο ζήτημα που αναφέρθηκε εδώ από τον Υπουργό και που καταγράφω ως επίτευγμα κοινό ε, Βελγίου, Ισπανίας και Ουγγρικής Προεδρίας, η οποία είχε όμως ίσονα ρόλο, διότι είχε πια σχεδόν κλείσει το θέμα όταν εμείς αναλάβαμε την Προεδρία. Εμείς μόνο την υπογραφή είχαμε να πραγματοποιήσουμε το Φεβρουάριο της Προεδρίας μας. Πάντως αποτελεί ορόσημο στη δημοκρατική ε, εμπλοκή των πολιτών στη δικασία λήψεων των αποφάσεων. Και έτσι, και έτσι έχει τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός, η εφαρμογή του, του αρχίζει σε ένα χρόνο από το, σημείο, από το η χρονική στιγμή της δημοσίευσης, δηλαδή από 1η Απριλίου του 2012 τίθεται σε εφαρμογή. Και είναι πιστεύω πολύ χρήσιμο και σημαντικό το μέσον αυτό που προσφέρεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης των θεμελιδών δικαιωμάτων. Προέβημεν σε μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής του χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων. Διατυπώσαμε σαφέστατη δέσμευση στον σεβασμό των θεμελιδών δικαιωμάτων και λάβαμε την έκθεση σχετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επί τη βάση της οποίας εκθέσεως ε, προέβημεν στην αξιολόγηση της υλοποίησης, ε, της εφαρμογής των όρων της χάρτας, του χάρτη μάλλον σε πεδίο Συμβουλίου αλλά και κρατών μελών και στις 23 Μαΐου στο Συμβούλιο υιοθετήθηκε ε, το σύνολο αυτών των συμπερασμάτων και πιστεύω ότι θα πρέπει κάθε χρόνο τακτικά πλέον το Συμβούλιο να προβαίνει σε μια τέτοια αξιολόγηση. Τη εφαρμογή του χάρτη. Η, Ευρω... η προσχώρηση Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Σύμφωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν μια από τι προτεραιότητε μα, το γνωρίζετε αυτό. Τι διαπραγματεύσει ξεκίνησε τις ξεκίνησε το προηγούμενο καλοκαίρι η Βελγική Προεδρία. Έχουν, έχουν γίνει ήδη, έχουν διεξαχθεί τρει διαφορετικοί γύροι διαπραγματεύσεων υπό την Ουγγρική Προεδρία. Ο προσεχή προβλέπεται για τι 20 με 21 με 24 Ιουνίου σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Σημαντικά βήματα όμω, και έτσι ήταν σε επίπεδο μόνο εμπειρογνωμόνων, σημαντικά βήματα έχουν επιτευχθεί στην υπόθεση αυτή και το καταγράφω επίση τη επιτυχία τη Προεδρία μα, χάρη και στι κοινέ προσπάθειε και την εξαίρετη συνεργασία μεταξύ ημών Επιτροπή και Κοινοβουλίου. Και το Κοινοβούλιο πρέπει να πω ότι είχε ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει τη διαδικασία αυτή. σε συνεργασία και με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί διεξήγαγε τις διαπραγματεύσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Φερρυπίν για την επιλογή ε, δικαστή. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εγγραφεί στις διαπραγματεύσεις. Όταν έρθει η ώρα, πιστεύω, θα αποδείξετε την στράτευση στην υπόθεση αυτή. Και αν μου επιτρέπετε τώρα, θα ήθελα να περάσω στα οριζόντια ζητήματα που αφορούν ε, τη σχέση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Όταν ορίσαμε το πρόγραμμά μας, τις προτεραιότητές μας, ιδιαίτερα εμείς είχαμε δώσει έμφαση ε, στην ενίσχυση της Ευρώπης ε, και με επίκεντρο τον πολίτη. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι είχαν πολλές δυσκολίες οι διοργανικές σχέσεις Φερρυπίν πολύ δύσκολες συζητήσει πέρσι το φθινόπωρο το χειμώνα εν του προϋπολογισμού και έτσι, μια και δεν φοβόμαστε τέτοιες μεγάλες προκλήσεις, αποφασίσαμε να διευκολύνουμε, να βελτιώσουμε αυτές οι οργανικές σχέσεις. Γνωρίζουμε, εξ αρχής γνωρίζαμε ποιες είναι οι δυσκολίες που θα είχαμε μπροστά μας. Μάλιστα κάποιοι προσπάθησαν και να μας αποθαρρύνουν ακόμα. Πιστεύω όμως Και το είδαμε και πολλέ φορέ όταν θέλησαμε να κερδίσουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε νομοθετικά θέματα, ότι μπορεί να είχαμε συμφωνία επί τη ουσία, αλλά στι διοργανικέ ε, συζητήσει, είτε να υπάρχουν προβλήματα επικοινωνία είτε διαφορετικές διαφορετικέ ερμηνείε, αποκλίνουσε ερμηνείε τη συνθήκη και έτσι να μην καταλήγουμε σε κοινό αποτέλεσμα. Πάντω, σαφέ είναι το εξή, ότι ο Ευρωπαίο ο πολίτη εν γέννη, δεν ενδιαφέρεται αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, επιμέρου θέμα στους πίνακες αντιστήξης, επί παραδείγματι, ή στο κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει απευθείας, ε, θα πρέπει να υπάρχει απευθείας νομοθέτηση, νομοθετική πράξη ή κατεχώρηση πράξη, του άλλους ο πολίτης δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν και τι συνεπάγονται αυτοί οι όροι. Ο πολίτης θέλει να μας βλέπει να λαμβάνουμε αποφάσει ουσιαστικέ. Άρα θελήσαμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα και με αυτό το πνεύμα ξεκίνησαμε τι διαπραγματεύσει και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο όρισε τη διαπραγματευτική του ομάδα υπό τον κύριο Ρέινεν και αρχίσαμε να επεξεργαζόμαστε διάφορα τρία διαφορετικά θέματα, του πίνακε αντιστοίχηση, τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι διεθνεί διασκέψει και την πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Με το Κοινοβούλιο λοιπόν συμφωνήσαμε ότι αυτά θα είναι τα τρία θέματα ζωτική σημασία. Αυτά τα θέματα δηλαδή τα οποία εντοπίζουμε ω εμπόδια στην πρόοδό μα σε ουσιώδη ζητήματα. Και επίσης συμφωνήσαμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας επιφέρει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την ε, συμμετοχή Φερρυπίν του Κοινοβουλίου σε διεθνείς διασκέψεις και άρα θα πρέπει να διευκολύνουμε και να κάνουμε τη σχετική προσαρμογή στη λειτουργία μας δεδομένου του ενισχυμένου ρόλου του Κοινοβουλίου. Ξεκίνησα από πλευρά μας λοιπόν τη δουλειά, σκληρή δουλειά σε επίπεδο Συμβουλίου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί συμφωνία από πλευρά Συμβουλίου στον τρόπο με τον οποίο μπορεί το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο Ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα μεγάλο, για ένα ζήτημα ευρύτατο, το οποίο θα προσδιορίσει και την πολιτική ατζέντα για τα επόμενα δύο χρόνια και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Φυσικά δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, είναι ενισχυμένο ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Και έτσι θέλαμε να έχουμε μια σαφή διαδικασία έτσι ώστε όταν η Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου καταθέσει την πρότασή της, τη νέα πρότασή της, να ξεκινήσει δουλειά αμέσως να μπορείτε να ανασκουμποθείτε και να πιάσετε δουλειά χωρίς να χιάνετε πολύτιμος χρόνος σε συζητήσεις για τα διαδικαστικά θέματα. Ύστερα λοιπόν από μακρές και δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών έχουμε καταλήξει μια συμφωνία και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να εξηγήσω για να αφήσω και το χρόνο για τις ερωτήσεις ε, τα επιμέρους ζητήματα Πρόσβαση στα απόρριτα στοιχεία λοιπόν, από τις πληροφορίες και πάλι από την αρχή της Προεδρίας μας ε, θεωρήσαμε ότι είναι πήγον το θέμα αυτό έτσι στο Κοινοβούλιο να έχει δυνατότητα πρόσβαση ε, στους φακέλους περί ε, πρόσβασης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο Σέγγεν για το οποίο είχατε και την ψηφοφορία, για το οποίο όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών έλαβε το Συμβούλιο πολύ σημαντικέ αποφάσεις. Δεν ήταν εύκολο μένα, αλλά καταφέραμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν την πρόσβαση για το Κοινοβούλιο στα έγγραφα αυτά. Μπορεί να μην αρκούν όμω αυτά. και χρειάζεται να βρούμε μια γενική λύση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ορίσουμε εμπειρογνώμονες για να δώσουν τις πρακτικές απαντήσεις για ε, να επιτευχθεί η συμφωνία. Το Συμβούλιο, που ξέρετε, έχει πολύ, πολύ αυστηρούς ε, κανόνες στο θέμα αυτό. το Κοινοβούλιο πιστεύω θα μπορέσει να, ορίσει, να εξασφαλίσει όρους ασφάλειας ε, το, για τα έγγραφα αυτά τα απόρριτα, αντίστοιχους με αυτούς που ισχύουν στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορούμε να αποδεσμεύσουμε, να αποχαρακτηρίσουμε απόρριτα έγγραφα για να έχετε και εσείς την πρόσβαση σε αυτά. Εκκρεμεί ένα ζήτημα οι προδιαγραφέ σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορέ μεταξύ ε, τη σχετική νομοθεσία των κρατών μελών ε, για ορισμένου βουλευτέ μπορεί να ισχύει αυτό για ορισμένου άλλου, να μην ισχύουν δηλαδή σχετικέ διατάξει στα κράτη-μέλη του. Άρα χρειάζεται να βρούμε μια κοινή λύση, μια λύση που να ισχύει για του πάντε και πιστεύω ότι στι διαπραγματεύσει αυτέ μπορούμε και κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας να δούμε την εξέλιξη εκείνη που θα φέρει σε αισιότερα στην υπόθεση αυτή. Για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε διεθνείς διασκέψεις, Το Συμβούλιο ήρε την ε, απέτηση για προηγούμενη έγκριση από πλευρά του Συμβουλίου και αποφάσισε την ε, έγκαιρη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με, ε, και, και αποφάσισε να μην απαιτεί όπω ορίζουν οι διατάξεις ε, πολύ προώρη ενημέρωση για το ποιοι βουλευτέ θα συμμετέχουν από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή να μην απαιτεί την ε, προειδοποίηση κατά τέσσερι εβδομάδες, αλλά μόνο δύο εβδομάδες για τα ονόματα των Ευρωβουλευτών και επιπλέον να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για εσωτερικέ συνεδριάσεις συντονισμού, ε, ώστε να, μπορεί το Κοινοβούλιο να παρακολουθεί μια υπόθεση και ταυτόχρονα το, Συμβούλιο να ε, λαμβάνει υπόψη και τι προτάσει ή τι παρατηρήσει του Κοινοβουλίου. Αυτή η διαπραγμάτευση έχει προχωρήσει, έχουν ήδη γίνει δύο γύροι. Ενημέρωσα την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο τον κύριο Λίνε και την ε, επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Μήνυ Ολομέλειας εδώ στις Βρυξέλλες θα ενημερώσω τη διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου για τις εξελίξεις ώστε να γνωρίζουν τι ε, φρονεί η Προεδρία για τους πινέκες αντιστοίχησης που αποτελούν πιστεύω το πιο δύσκολο θέμα αυτό που μας εμποδίζει από την πρόοδο στην νομοθεσία η κατάσταση έχει ως εξής Υπάρχει η διοργανική συμφωνία του 2003 μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, η οποία ορίζει ότι η χρήση πινάκων αντιστοίχησης θα πρέπει να ενισχύεται. Εν τω μεταξύ, τον προηγούμενο Δεκέμβρη, η διάσκεψη των Πρόεδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιφάσισε ότι δεν μπορεί να υιοθετείται οδηγία από το Κοινοβούλιο στη διαδικασία της συναπόφασης εάν δεν συμπεριλαμβάνει και πίνακες αντιστοίχησης Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν πως είναι υποχρεωτική η χρήση των πινάκων αντιστοίχησης. Έκτοτε δυσχέρανε ιδιαίτερα η νομοπαραγωγική διαδικασία. Διότι το Συμβούλιο δεν συμμετέσχει σε αυτή τη συμφωνία και τα κράτη-μέλη δεν δέχονται να λαμβάνει αποφάσεις στο Κοινοβούλιο που τους επιβάλλουν μια υποχρέωση χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Ξεκινήσαμε τι διαπραγματεύσει με την ε, τρέχουσα διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου. Έχουμε κάνει δύο προτάσει εκ μέρου των κρατών μελών, μάλλον για τα, προ τα κράτη-μέλη. Δεν τι δέχθηκαν τα κράτη-μέλη. Ε, συνεργαζόμαστε με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή. Αλλά προσκρούμε στο γεγονό ότι θέλησε το Κοινοβούλιο να καταστήσει υποχρεωτικού του πίνακε αντιστήξεις. Αυτό δυσκολεύει πολύ τη ε, δουλειά μα γιατί δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο είναι, αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τα κράτη-μέλη για μια συμβαστική κίνηση που θα οδηγούσε στην επίλυση του ζητήματο. Εμεί κάναμε πολύ συγκεκριμένε προτάσει. και σε ορισμένα στάδια της διαπραγμάτευσης είχα την εντύπωση όπως και όταν ήμουν παρούσα στη διάσκεψη των Προέδρων, είχα την εντύπωση ότι υπήρχαν ε, τάσεις από πλευράς των Ευρωβουλευτών να ακολουθήσουν την πρόταση της Προεδρίας, ότι λέει, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε πιο πολύ στην ουσία και όχι στα ε, θεσμικά ζητήματα ή στα θέματα της οργανικής συνεργασίας. Ε, και μπορέσαμε σε ορισμένα σημεία να προχωρήσουμε περισσότερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η εξέβρεση ενός γενικού μόντους βιβέντη, προκειμένου να βγούμε από αυτό το διέξοδο. Κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Φερρυπίν, χρήση των ε, πινάκων αντιστοίχησης για τον εμβολιασμό των ε, αγελάδων σε περίπτωση αυτόδους πυρετού. Ε, αλλά από την άλλη Πώ μπορεί κανεί να εξηγήσει τον πολίτη ότι δεν θα γίνει εμβολιασμό τη Αγελάδα όταν έχει ενσκέψει μια τέτοια επιδημία, μόνο και μόνο επειδή δεν συμφωνούν τα δύο θεσμικά όργανα για το σπίναξ τη τύχηση. Επίση, προτείνουμε, και αυτό προκύπτει και από τι διαπραγματεύσει, ένα μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεις έκανε την πρόταση το κοινοβούλιο να ε, προχωρήσει σε άρση τη εφαρμογή αυτής τη απόφασης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει το Συμβούλιο να έχει ένα περιθώριο για εξέβρεση μια συμβαστική λύση, δηλαδή να βελτιωθεί το κλίμα λίγο πολύ. Και έτσι τα θέματα τα οποία έχουν ε, βαλτώσει λόγω του προβλήματος των πινάκων αντιστοίχησης να μπορέσουν να προχωρήσουν σε έγκριση και να κερδίσουμε ένα περιθώριο χρονικό, φερρυπίν, για το θέμα του εμβολιασμού. Αυτή η πρόταση λοιπόν για μια περίοδο χάριτος απερίφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα μια νέα πρόταση. Απάντηση δεν έχουμε λάβει ακόμη. Δηλαδή, εμεί απλώ συνοψίσαμε ποια είναι τα θέματα που παραμένουν εκκρεμοί λόγω των διοργανικών αυτών προβλημάτων, είτε πρόκειται για την ε, εκτελεστική πράξη της κατεχώρηση ε, πράξης, είτε για τους πίνακες αντιστοίχησης. Έχω εδώ ένα κατάλογο για όποιον ενδιαφέρεται. Καταγράφουμε λοιπόν τα σημεία που παραμένουν εκκρεμή, στα οποία έχουμε εξεύρει συμφωνία επί της ουσίας και προσκρούμε μόνο σε νομικά ζητήματα και όπου πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στον πολίτη, Φιρυπίν, στους φοιτητές από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ότι δεν μπορούν να ε, λάβουν τις υποτροφίες ε, που δικαιούνται γιατί εμείς μεταξύ μας δεν τα βρίσκουμε. Εάν πρόκειται δηλαδή για κατεχώρηση ε, πράξη, για απευθείας νομοθετική πράξη και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά ζητήματα. Έχουμε πολλούς και πολλά ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή εδώ και μήνες λόγω αυτών των διοργανικών σχέσεων. Το ίδιο και για τους μπάνανο παραγωγούς που δεν μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους λόγω αυτών των διοργανικών προβλημάτων. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εδώ περισσότερη ευελιξία θα ήταν χρήσιμη και για μας. Όπως επίσης θεωρώ ότι έχουν και τα δύο θεσμικά όργανα ευθύνη, το Συμβούλιο και το, και το Κοινοβούλιο, ε, να προχωρήσουν σε συμφωνία. Να εξασφαλιστεί πρόοδος δηλαδή τα θέματα αυτά. Σταματώ εδώ μακρηγόρησα και ζητώ συγγνώμη, αλλά ήθελα να σας δώσω το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα αυτών των διοργανικών θεμάτων. Ένα θέμα ακόμη μόνο, μου επιτρέπετε, για το Μητρό Διαφάνειας, που είναι πολύ σημαντικό για σας, πιστεύω, και όπου εγκρίνατε και ένα ψήφισμα. Μάλιστα στις σχετικές συζητήσει ε, είχα λάβει και εγώ το λόγο. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι έχει υπογραφεί η διοργανική συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Και μετά τις προσπάθειες που κατέβαλε και η Προεδρία μας δόθηκε η άδεια να λέμε ότι όταν υπογράφεται μια διοργανική συμφωνία πρέπει να κάνουμε πολιτική δήλωση προς το Συμβούλιο είναι έτοιμο και διατεθειμένο να προχωρήσει σε ε, τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το ρόλο και τις ετυπώσεις συμμετοχή του Συμβουλίου σε αυτό το Μητρό Διαφάνειας. Βέβαια, ο ρόλος μας είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του, Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, γιατί εμείς ως θεσμικό όργανο δεν είμαστε εκτεθειμένοι στις πιέσεις των ομάδων συμφερόντων. Είναι ίσως η κυβέρνηση των κρατών μέλων, αλλά πάντως όχι εμείς ως θεσμικό όργανο. Και άρα έχει άλλη βαρύτητα η δική μα συμμετοχή. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία το ότι θα συμβάλλει σε αυτό το θέμα τη διαφάνεια, του Μητρώου Διαφάνεια, στο Κοινοβούλιο. Και επίση στη διαδικασία που θα μπορούσε να επιτρέψει την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, Απέστειλε ο πρόεδρός μας ε, επιστολή στον πρόεδρο Μπούζεκ την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία του εγχείρησα εγώ μάλιστα, για τις συζητήσεις ε, σε επίπεδο προέδρων αλλά και ε, εκπροσώπων του Κοινοβουλίου με την πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου, επαφές με την Προεδρία και στο επερχόμενο, στην επερχόμενη Τρόικα ή Τρίο, έτσι ώστε να λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σας όπως θέλετε σωστά και θα είμαστε στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω. Ελπίζουμε την πρόταση αυτή της Προεδρίας μας να την κάνει δεκτή το Κοινοβούλιο. Την ε, υποστηρίζει άλλωστε και η τριανδρία των επόμενων Προεδριών και η Επιτροπή από ό,τι ξέρω. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά είχα να σας πω για τα θέματα των αρμοδιοτήτων μας, σας, της Επιτροπής σας. Ήθελα να σημειώσω ότι ήταν ε, πολύ ευχάριστη η συνεργασία μας σε όλους αυτούς τους μήνες. Παραδίδουμε τη σκητάλη της Προεδρίας στο Συμβούλιο ΜΕΝ. Ελπίζω όμως ότι θα επικρατήσει και κατά την επερχόμενη Προεδρία αυτή η θετική προς το Κοινοβούλιο στάση. Και πάντως σας διαβεβαιώνω ότι η Ουγγαρία από εδώ και μπρος ακολουθεί μια φιλική για το Κοινοβούλιο στάση, όχι πλέον ως Προεδρία, αλλά ω κράτος μέλο. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριε Γιώργη για μια αναλυτική παρουσίαση. Θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου. Θα ήθελα να πω ότι εγώ ασχολήθηκα με το θέμα του, της διαφάνειας ε, ε, του Μητρώου Διαφάνειας λοιπόν Νομίζω ότι και σε πρακτικό επίπεδο πολλά μένουν να ρυθμιστούν, αλλά δεν θα πρέπει να εξαιρέσει κανείς, να αποκλείσει κανείς ότι μπορεί να υπάρξουν πιέσεις από πλευράς κρατών μελών, από πλευράς μελών του Συμβουλίου κτλ. Νομίζω ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα συμφωνήσει με αυτό το Μητρό Ασφαλείας, αυτό θα έχει μια σημασία ιδιαίτερα συμβολική γιατί θα δείχνει την διαφάνεια του συνόλου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει, θα πρέπει λοιπόν και το Συμβούλιο <clears throat> ως εκπρόσωπος των κρατών μαζί με το Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος των λαών της Ευρώπης να μπορέσουν να συνεργαστούν σωστά σε ένα πλήρες καθιστός ε, διαφάνειας. Η Ουγγαρία γενικά υποστηρίζει τις θέσεις του Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας. Η κυρία Τσίτα Γκούρμα έχει ζητήσει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή κυρία Γκέρι, ε, τα τέλη, ε, Ιανουαρίου ε, μίλησε σε εμάς ο κύριος Μαρτίνη και νομίζω ότι πραγματικά αναφέρθηκε σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. ανέφερε όλα όσα θα ήσαν σημαντικά στο πλαίσιο της Ουγγρικής Προεδρίας. Παρουσίασε επίσης ορισμένα πακέτα τα οποία θα ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και ε, επίσης υπήρξαν ορισμένα συνταγματικά θέματα, η αλλαγή της συνθήκης ή και κάποια άλλα ζητήματα και επίσης επισημάνθηκε ότι πραγματικά πολλά είναι κατεπήγοντα θέματα που θα πρέπει να εφαρμοστούν τάχιστα. Ορισμένα πέτυχαν, αλλά όχι. Άλλωστε τα είπατε και η ίδια, κυρία Υπουργέ αλλά σας χαίρομαι πάρα πολύ που μας επισημάνατε ότι πρωτοβουλίες, η πρωτοβουλία των πολιτών ε, κατέληξε σε επιτυχία και εγώ ήμουν υπεύθυνη εδώ εκ μέρους της Επιτροπής ε, ΑΦΚΟ και νομίζω ότι και εγώ μπόρεσα να συμβάλλω θετικά. Επίση, η προσχώρηση τη Κροατία υπήρξε ένα ιδιαίτερο σημαντικό θέμα για την Ουγγρική Προεδρία και στις 24 ε, και 25 του μηνός θα υπάρξει μια συνάντηση κορυφής εδώ στις Βρυξέλλες και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραφούν τα κείμενα αυτά, γιατί αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό για πολλούς εξημών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια αυτή. Τώρα το Europlus ε, πρόκειται για μια προσθήκη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, πρόκειται για ένα θέμα της κοινή οικονομικής πολιτικής και της κοινή οικονομικής διακυβέρνησης και είναι σημαντικό εδώ να ληφθούν υπόψη και οι στόχοι των επιμέρους χωρών μελών. Ε, τρία μέλη, κατά κάποιο τρόπο πηγαίνει το καθένα στο το δικό του δρόμο. Θα πρέπει κάπως να συντονιστούν οι προσπάθειες και να ενισχύσουμε και την σταθερότητα του νομίσματός μας. Αυτό είναι ένα σημαντικός, αυτός είναι ένα σημαντικός στόχος και εδώ υπήρξαν σημαντικές ε, αντιστάσεις. Τώρα, πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα με το Σέγγεν. Και εδώ έγινε μια ζωηρή συζήτηση. Επίσης το θέμα της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ε, νομίζω ότι πραγματικά ήταν ένα από τα πιο σημαντικά εγχειρήματα κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας και ε, έγινε και μια συνεδρίαση στην Βουδαπέστη σχετικά με το θέμα αυτό. Επίσης το ζήτημα της ε, χρηματοδότησης και ποια, θα είναι, ποια, διαφαίνε, ποια εξέλιξη διαφαίνεται. Αυτό το θέμα ίσως κάπως μπήκε στην άκρη, αλλά έχω πιστοσύνη ότι θα μπορέσει να επιτευχθεί μια συμφωνία με την ε, Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και μας παρουσιάσετε τα αποτελέσματα πραγμένα της Ουγγρικής Προεδρίας. Σίγουρα τα πράγματα δεν ήταν εύκολο, αλλά συνολικά νομίζω η εντύπωση που σημάτισα είναι ότι πραγματικά ήταν, υπήρξε τετέρως επαγγελματικό το έργο σας. Μετά την παρέμβαση της κυρίας Γκορμάη έχει ζητήσει το λόγο ο συνάδελφος Πρόντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε την εφαρμογή του, της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όπως ξέρετε, τις χώρες, μαζί και η Μεγάλη Βρετανία, ε, σας δόθηκε ένα opt-out από τη Χάρτα. Ε, επίσης, για την Τσεχία ήταν το τίμημα που πλήρωσαν για την υπογραφή της Εθήκης της Λισαβόνας ορισμένα μέλη αυτής της Επιτροπής που γνωρίζει περισσότερα για συνταγματικά θέματα μου είπαν ότι αυτά τα opt-out είναι άχρηστα γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας που βλέπει μια υποχρέωση εφαρμογής. Ε, ορισμένα μέλη της Επιτροπής και εκπρόσωποι της ε, Προεδρίας και άλλοι ε, ειδικοί σε συνταγματικά θέματα αρνήθηκαν να δεν μου έδωσαν μια ικανοποιητική απάντηση ενδεχομένως ε, υπάρχει μία αντίδραση στις χώρες ε, μέλη και μπορεί να, δοθεί, να γίνει τελικά ένα opt-out μέσω μιας διαφορετικής οδού. Αυτό το οποίο ζητώ είναι τα ζητήματα της ε, εφαρμογής της χάρτας και της δυνατότητας του opt-out. Είναι ισχύει αυτό το δικαίωμα ή είναι εντελώς άχρηστο όπως υπόθηκε. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Ε, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ ευχάριστο που σας βλέπουμε εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους των, της των φιλελευθέρων για την σκληρή ε, εργασία. Αλλά υπάρχει, έχω την αίσθηση κάποια απογοήτευση για το ότι δεν μπορέσετε να κάνετε περισσότερα πράγματα κατά τη Προεδρία σα. Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλε τι Προεδρίε. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αυτό να το μια διάκριση εναντίον σα. Ε, έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μια αντίδραση στην συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς ε, οι πολίτες ε, αρχίζουν να κατανοούν την πλήρη εμβέλεια της συνθήκης. Όπως είπε ο κ. Μπρόνς, στη χάρτα ε, δεν ε, τίθεται θέμα του να, να έχει η Μεγάλη Βρετανία το δικαίωμα του opt-out. Δεν μπορεί να το πράξει πράγματι. Το πρωτόκολλο περιορίζει την ε, ελευθερία των Βρετανικών δικαστηρίων όσον αφορά κάποιες ε, διενέξεις και δεν μπορούν οι Βρετανοί πολίτες κατά συνέπεια να έχουν την ε, πλήρη προστασία της ε, χάρτας στην περίπτωση αυτή. Η Βρετανική κυβέρνηση είναι αυτή η οποία μιλάει για ένα δικαίωμα opt-out και νομίζω ότι αυτό είναι κάπως παραπλανητικό, κύριε Πρόντσο. Όσον αφορά τους πίνακες αντιστοίχησης, είναι σαφές ότι πραγματικά μπορεί να, ε, να μας γίνει μια ειδωληψία το ζήτημα αυτό των πινάκων. Ε, βέβαια χρειάζεται κάποια ευελιξία εδώ και αυτό το ζητάει και το Συμβούλιο. Ο λόγος που θέλουμε αυτούς τους πίνακες είναι, είναι επειδή πιστεύουν ότι αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας ε, και τις διαφάνειας επίσης. Και νομίζω ότι οι χώρες ε, μέλη αποφασίζουν ε, τι τους χρειάζεται για να εφαρμόσουν τον ευρωπαϊκό νόμο, να το μεταγράψουν σε εθνικό νόμο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα δράσης. Και θεωρώ ότι αυτό αφορά ορισμένους από τους συναδέλφους στο Συμβούλιο που πραγματικά έδειξαν ιδιαίτερο πείσμα, επέμεναν ιδιαίτερος στο να εμποδίσουν, να παρεμποδίσουν την ε, ροή της νομοθεσίας. Ε, μπορείτε να είστε πιο ακριβείς όσον αφορά τις συζητήσεις και τις συμφωνίες για το πολιτές πλαίσιο και να μας πείτε κάποια πράγματα για την ε, διασύνδεση με τις διαπραγματεύσεις για το MFF από τη μία και το ζήτημα των πόρων από την άλλη. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια περιεκτική συνολική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Επίσης πιστεύω ότι το αίτημα του Κοινοβουλίου να γίνει μια διακοινοβουλευτική ε, για να ανοίξουν τα ζητήματα αυτά, όχι μόνο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, όχι μόνο όσον αφορά τις επιτροπές προϋπολογισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά αυτές που ασχολούνται με την, ε, με αξιοποίηση των κονδυλίων. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία επ' αυτού, εάν δεν έχουμε μια πλατιά, ένα πλατή και βάθος προβληματισμό που να περιλαμβάνει όλα τα κοινοβούλια. Αν η διαπραγμάτευση περιοριστεί μόνο στους ε, Υπουργούς Οικονομικών δεν θα υπάρξει συμφωνία και θα ε, καταδικαστούμε τελικά να ε, παραμείνουμε στις παρούσες προοπτικές και αυτό θα ήταν ολέθριο. Όσον αφορά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα σχέση με τα 18 μέλη, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Well, Minister, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Νομίζω ότι πράγματι νιώσαμε ότι ήσασταν μια Προεδρία φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφερθήκατε και σε κάποια εύκολα θέματα, τα οποία δεν χρειάζεται πολύ πολιτικό θάρρος, σχετικά με το Δελτανιτάφ σαν παράδειγμα και για τους ε, πίνακες αντιστοιχίας και γι' αυτό θα ήθελα να σας θέσω και άλλες εύκολες ερωτήσεις η μία αφορά, ξέρω ότι θα απαντήσετε με διπλωματία βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να δώσετε διαφορετικού τύπου απαντήσεις. Οι σχέσεις ανάμεσα στις Εθνικές Προεδρίες και στη Μόνιμη Προεδρία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σίγουρα θα πρέπει να δείξετε μια κάποια διπλωματία στην απάντηση. Αλλά αν ένα πράγμα θέλετε να βελτιώσετε στις σχέσεις ανάμεσα στις εναλλασσόμενες προεδρίες και τη μόνιμη προεδρία, ποιο θα είναι. Επίσης η απουσία, ε, εν πάση περιπτώσει, από συζητήσεις που γίνονται για τα θέματα της ΚΕΠΑ είναι κάτι το οποίο εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι σημαντικό ή πιστεύετε ότι η δουλειά την οποία έκανε η, προ, μόνιμη Προεδρία ε, δεν απαιτούσε και τη δική σας παρουσία. Πριν έρθετε εδώ συζητήσαμε και το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις δικές σας εκτιμήσεις για τις διαπραγματεύσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ιδιαίτερα σχετικά με τις απαιτήσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την συνέχεια της διαδικασίας. σχετικά με τις μόνιμες και διαφανείς ε, διαδικασίες γύρω από το θέμα των προμηθειών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα επίση να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία με την Ουγγρική Προεδρία. Αλλά θα με ενδιέφερε να έχουμε και μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων γιατί η Προεδρία σας πραγματικά αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες όχι μόνο λόγω της παρούσας κρίσης, αλλά λόγω των προβλημάτων σε σχέση με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και των σχέσεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή. Σε ποια κατεύθυνση θα πάνε τα πράγματα και κατά πόσο ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και σε μια επικοδομητική συνεργασία ή κατά πόσο, είμαστε, ε, κατά πόσο δεν είμαστε σε θέση να το πράξουμε. Ε, εδώ παίζει ένα ρόλο η σχέση με τα εθνικά κοινοβουλία και όλο το πλέγμα των θεσμικών οργάνων, των εθνικών και των ευρωπαϊκών. Ε, όλα αυτά στέκονται πάνω σε πύληνα πόδια, γιατί δεν υπάρχει μια ομοφωνία εδώ, μια ενότητα. Και πραγματικά μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται για να μην ξεσπάσει ένας θεσμικός πόλεμος. Έχω την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο αγωνίζεται για τα δικαιώματά του αλλά ορισμένες φορές υπάρχουν κάποιες αμυντικές αντιδράσεις ή αμυντικά αντανακλαστικά εκ μέρους του Συμβουλίου, όπως γίνεται με την Κορεπέρ όπου πραγματικά γίνονται πάρα πολλές ε, υπερβολές, οι ενδράσεις εδώ είναι υπερβολικές. Και μπορώ να φανταστώ ότι εδώ μέσα σε αυτό το πλέγμα ε, μία δυσκολία για σας στο επίπεδο της Προεδρίας ήταν να διαπραγματευτείτε συνδυασμούς με το Κοινοβούλιο ε, από την άλλη ε, να μπορέσετε ε, να έχετε διαπραγματιστική να διατηρήσετε μια διαπραγματευτική ικανότητα, η ισχύ. οι διπλωμάτες προσπαθούν να κρατήσουν τα ενία, κάτι που τους φέρνει ακόμα τα πράγματα. Ελπίζω παρόλα αυτά ότι θα μπορέσουν να βρεθούν κάποιες λύσεις. Επιτρέψατε μου να, σας, να πω κάτι σε σχέση με τα όσα είπε ο Βρετανός συνάδελφος για τη Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Το ζήτημα αυτό δείχνει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει διαβάσει τη Χάρτα των Θεμελιδών Δικαιωμάτων η οποία απευθύνεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και γι' αυτό το λόγο ε, ε, απευθύνεται μόνο σε αυτά τα θέματα. Ως εκ τούτου ε, δεν είναι δυνατόν ε, να υπάρξει εθνική παρεμβολή. Αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δικαιολογημένα η Μεγάλη Βρετανία ε, ζήτησε ένα opt-out για κάτι για το οποίο έχουν opt-out ούτως ή άλλως όλες οι χώρες μέλη γιατί δεν πρόκειται για εθνική νομοθεσία όπως σας είπα. Και έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Γκαλτιέρη. Ευχαριστώ Υπουργέ. Και εγώ θα συμφωνήσω για τα ευχαριστήρια στα οποία αναφερθήκατε θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπροκ και στην δυσκολία την οποία αντιμετώπισε η Προεδρία σας στα πλαίσια μιας φάσης η οποία μας επιβάλλει να αντιμετωπίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο βαθύτατα ανανεωμένο μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, συνειδητοποιώντα ταυτόχρονα τις επιθυμίες που έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες αυτές. Το θέμα δεν είναι μόνο λοιπόν η εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της νέας συνθήκης, αλλά η αφομοίωση θα έλεγα επί της ουσίας αυτής της ειρηνικής επανάστασης μετά το τέλος του καθεστώτος των πυλώνων και με τον ορισμό πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως άμεσου εκπροσώπου των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αυτές τις αλλαγές ε, θα υπάρξουν συνέπειες όπως επίσης και από άλλες αλλαγές όπως το θέμα της μόνιμης προεδρίας κτλ. Δημιουργούνται λοιπόν ορισμένες τριβές πλέον οι τριβές αυτές ίσως ε, προέρχονται και από την αδυναμία μας, από την κόποση απορρόφησης αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου. Και γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στις εμπειρίες τις οποίες εσείς βιώσατε. Ε, μία ερώτηση πρώτη λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εσείς πειραματιστήκατε και ζήσατε μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εμείς εδώ και λίγη ώρα συζητήσαμε την περίεργη φύση ενός, ενός εξαμήνου ευρωπαϊκού χωρίς νομική βάση που βασίζεται στην αναθεώρηση ενός κώδικα συμπεριφοράς. Αλλά τεχνικά δεν υπάρχει το, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Βέβαια, επί της ουσίας υπάρχει. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν την ανάγκη να προσδώσουμε μια κατάλληλη νομική βάση στο ευρωπαϊκό εξάμεινο επί του 121.6 του κανονισμού που θα επιτρέψει το να καταστήσουμε το εξάμεινο αυτό το σταυροδρόμι του συνόλου των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο του Συμφώνου Σταθερότητας. Το δεύτερο θέμα αφορά τις καινοτομίες τις οποίες εισάγει η συνθήκη στις διεθνείς συμφωνίες που και αυτό έχει τεθεί για συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο. Θα ήθελα να πω και σαν μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας και Ασφάλειας ότι δεν υπάρχει μια σαφής κατανόηση του καινοτόμου το οποίο προτείνεται από το 118 που αποκλείει από τη διαδικασία τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Μόνο τις διεθνείς συμφωνίες οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στην ΚΕΠΑ αποκλειστικά στην ΚΕΠΑ, όχι κυρίως ε, να εντάσσονται στην ΚΕΠΑ. Όποιες δεν είναι 100% ΚΕΠΑ απαιτούν την γνώμη και την ε, συνένεση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν παρόλα αυτά συμφωνίες οι οποίες έχουν ληφθεί με βάση νομική την ΚΕΠΑ όπως η τελευταία συμφωνία για τις εκδόσεις σε θέμα δικαστικό δηλαδή ε, τέθηκε και το θέμα της διαδικασίας Αταλάντα της αποστολής στην Ίσο Μαυρίκιο που ε, προχώρησε χωρίς να ακολουθηθεί κατάλληλη κατεμέ διαδικασία, κάτι το οποίο καθιστά τη συμφωνία αυτή για το Αταλάντα παράνομη. Συνεπώς, τι θα γίνει λοιπόν με το θέμα αυτό της αφομοίωσης των συνεπειών της νέας συνθήκης. Χέφνες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα, επί τη ευκαιρία, να επανέλθω σε ένα μόνο θέμα, γιατί τα παστορία έχουν καλυφθεί από τους συναδέλφους. Και έχει προχωρήσει και η ώρα. Το θέμα της πρωτοβουλίας των πολιτών. Γιατί σε μια προσωπική συζήτηση είχα επισημάνει ότι η έγκριση του θέματος τον Απριλίου ουσιαστικά δεν το κλείνει και ότι παραμένουν εκρεμή πολλά ζητήματα. Και έτσι έχουμε κάποιες ανησυχίες, διότι ενδέχεται σε ορισμένα κρατημέλη, σε αρκετά κρατημέλη, η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό ε, δίκαιο να προχωρήσει κατά τρόπον πολύ διαφορετικό από, μέλος, από κράτος σε κράτος. Μερικές φορές δεν είναι γνωστό καν ποια αρχή είναι αρμόδια ε, ή ορισμένα κράτη-μέλη μας επισημαίνουν ότι δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν όσο έχει τη διάταξη περί online υπογραφής στο, στο αίτημα αυτό, γιατί δεν έχουν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου που απαιτείται. Ε, άλλες κυβερνήσεις λένε ότι μπορεί να απαιτείται από τον κανονισμό το λεγόμενο random checks, δηλαδή τυχαίοι έλεγχοι, περιστασιακή έλεγχη, αλλά μπορεί να οδηγήσει η θέση σε εφαρμογή του συστήματος αυτού σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις από διοικητικής πλευράς. Ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι χρειάζεται σαφώς ε, συντονισμός από πλευράς του Συμβουλίου συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών ώστε να φτάσουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα, σε μια ενιαία δηλαδή, αλλά και εύχρηστη για τον πολίτη, ουσιαστική ε, εφαρμογή του συστήματος αυτού. Ήθελα να σας το επισημάνω. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες, ε, στις εβδομάδες που σας μένουν, να μπορέσετε να βελτιώσετε λίγο την εφαρμογή του σε σχέση με τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Έχετε πολλά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και τα όσα εκφράσατε εκτιμώντας το έργο της Προεδρίας. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το Μητρό Διαφάνειας, Είπα ήδη στις αγωγικές μου παρατηρήσει ότι ναι, πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό και χαιρετίζουμε τη δέσμευση αυτή που ανέλαβε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να πετύχουν μια συμφωνία όσον αφορά το Μητρό Διαφάνειας και την πολιτική δήλωση που θεωρώ ότι είναι θετικό βήμα εκ μέρους του Συμβουλίου. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε αυτή την εργασία και ε, συνεχή βάση θα, το, ε, θα κάνουμε αξιολογήσεις και θα λάβει μια σχετική απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, ευγενικέ σας παρατηρήσεις καθώς και τις ε, ειδικέ σας ε, και τις ειδικές ερωτήσεις. Θα υπάρξει ένας γύρος διαπραγματεύσεων στις 25 Ιουνίου θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό ούτω ώστε να δούμε τι γίνεται με όλα τα κεφάλαια της ε, διαπραγμάτευσης. Και εάν όλα πάνε καλά θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τέσσερα νέα κεφάλαια και θα κλείσουμε τα παλιά κεφάλαια γιατί μιλούμε για, για μια χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Συνεπώς υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν για παράδειγμα τις δημοσίες προμήθειες, την εκπαίδευση και ορισμένα άλλα κεφάλαια, την έρευνα για παράδειγμα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα ανοίξουμε όσον αφορά, και να κλείσουμε κάποια άλλα. Όσον αφορά το Schengen, ε, δημοσιοποιήθηκε η γερμανογαλλική ε, προεδρική επιστολή βάσει της οποίας ε, μάθαμε ότι δεν θα υπάρξει προσχώρηση κατά τη διάρκεια της, ε, προεδρίας, της, Βουλγα... της Ουγγρικής Προεδρίας ε, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Θα πρέπει να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που μας ε, παρήχαν. Νομίζω ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση εδώ την περασμένη εβδομάδα σημαντική δουλειά έγινε και ορισμένες χώρες ήταν κατά. Συγκεκριμένα 7 χώρες, οι οποίες όμως στη συνέχεια άλλαξαν τη γνώμη τους. Και τώρα γνωρίζουμε το πώς σκέφτονται αυτές οι χώρες και η Ιρμανία και η Βουλγαρία γνωρίζουν πώς σκέφτονται οι άλλες χώρες για αυτές. Γνωρίζουμε λοιπόν τις προσπάθειες που κάνουν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα εθνικά κριτήρια της προσχώρησης στο Σέγγεν έχουν εκπληρωθεί από αυτές τις δύο χώρες. Αυτή είναι μια τεράστια εξέλιξη, μια τεράστια επιτυχία και μας είπαν ότι το Σεπτέμβριο θα επανέλθουν στην απόφαση αυτή και θα ληφθούν αποφάσεις για μελλοντικά βήματα. Επίσης ε, ε, λέχθηκαν κάποια πράγματα για τον οδικό χάρτη και νομίζουμε ότι θα υπάρξει μια λύση. Οι πολιτικές αποφάσεις ελπίζουμε θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας και οι θέσεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων κατατείνουν προς μια σύγκληση και νομίζω ότι αυτό είναι μια, επιθυμ... Ε, είναι μια επιτυχία. Όσο για την συνάντηση ACP και την συνάντηση της ΚΟΖΑΚ, νομίζω ότι ήταν πολύ θεατική η συμβολή του στην Προεδρία. Ο Πρωθυπουργό έλαβε μέρο σε αυτή τη συνάντηση και υπήρξε ιδιαίτερη καρποφόρα συνάντηση ε, και συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τέθηκαν πάρα πολλές ερωτήσεις και ε, νομίζω ότι πραγματικά έχουμε κατά νου μια ισχυρή ευρωπαϊκή εκστρατεία. Ε, θα υπάρξει μια επιστολή απάντησης, αυτό είναι νομικό τεχνικό ζήτημα και έγινε μια εκστρατεία στην Ουγγαρία δεν αφορά τις ε, ρυθμίσεις για την έκτρωση που δεν άλλαξαν αλλά πρόκειται για τις ίσες ευκαιρίες εκ μέρους της Ουγγρικής κυβέρνησης. Θέλουμε να δώσουμε λοιπόν μια ευκαιρία προς εκείνους τους ε, γονείς που επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Και ε, όσον αφορά την έκδοση, αν πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το θέμα, οι γονείς αυτοί έχουν πιο περιορισμένες επιθυμίες, ε, δυνατότητες συγγνώμη, υιοθεσίες ενός παιδιού. Βεβαίω θα υπάρξει μια νομική και τεχνική συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν σχέση με το κατά πόσο όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προόδου ή όχι εάν ε, η έκβαση αυτής της συζήτησης ε, θα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό, τότε θα αντλήσουμε ορισμένα συμπεράσματα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα επίσης να σας πω το πώς σκέφτεται η Ουγγρική Προεδρία για το θέμα αυτά. Όσο για τον κύριο Μπρόντς, θα ήθελα να πω ότι η ερώτησή σας εν μέρη έχει απαντηθεί όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ήθελα να συνεχίσω στα αγγλικά. Όσον αφορά το δικαίωμα του opt-out από τη χάρτα, η Τσεχία είχε ζητήσει αυτό το δικαίωμα σε μια μεταγενέστερη φάση και ε, το Συμβούλιο είπε ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να τεθεί στην επόμενη τροποποίηση συνθήκης όταν ενταχθεί η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς λοιπόν το θέμα αυτό εκκρεμεί. Αλλά βέβαιο είναι ότι η χρονική συγκυρία είναι ξεκάθαρη, αλλά θα υπάρξει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό νομοθέτημα, γιατί ε, αφορά μια τροποποίηση της συνθήκης με την προσχώρηση μιας χώρας. Ελπίζω ότι θα υπογραφεί η συνθήκη. Είναι πολύ δύσκολη βέβαια η προετοιμασία του νομικού κειμένου της ε, προσχώρησης και ελπίζω ότι στην περίπτωση αυτή ε, θα βρεθεί μια καλή λύση για αυτή την επιπρόσθετη ε, τροποποίηση της συνθήκης εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Ευχαριστώ κύριε Τάφ. Στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι καμία απογοήτευση. Απλώς θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της αμοιβαίας μας ευθύνης για να είμαστε αποτελεσματικοί και να ασχολούμεθα με την ουσία. Γιατί νομίζω ότι αυτό απαιτούν από εμά οι πολίτε. Και ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονό ότι διαπιστώσαμε ότι όποτε συνεργαζόμαστε με του ε, εισηγητέ και τι διάφορε επιτροπέ, πάντοτε μπορέσαμε να βρούμε ένα μόντου βιβέντη. Ε, Όταν ε, το ντοσιέ αυτό πήγε σε ανώτερα πολιτικά στρώματα, ας το πούμε έτσι, τέθηκε το θέμα αυτό των πινάκων αντιστοίχησης, διοργανικής συνεργασίας κλπ. Και είναι ξεκάθαρο ότι οι εισαγητές στην περίπτωση αυτή βρέθηκαν σε μια ε, διαφορετική κατάσταση γιατί πάλευαν για, την, ε, για τις ιδέες τους και τελικά παρακολύονταν. Ε, θεωρώ ότι εμείς δώσαμε ξεκάθαρα μηνύματα και υποβάλαμε ξεκάθαρες προτάσεις που όταν διευκολύνουμε αυτή τη σχέση ελπίζουμε ότι θα ανταμυφθούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να κατανοήσει τα κίνητρά μας. Όσον αφορά τους ε, πίνακες αντιστοίχησης, συμφωνώ είναι καλό για τη διαφάνεια. Η δική μου χώρα μέλος, που είναι καινούριο μέλος, ε, ε, εδώ είχαμε πάντοτε την πρακτική αυτή. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτούς τους πίνακες αλλά κατανοώ ότι σε σχέση με άλλα μέλη μπορούν να ανακύψουν κάποια προβλήματα, ιδιαίτερως για εκείνα τα μέλη που έχουν ομοσπονδιακή δομή, για παράδειγμα όταν γίνεται η μεταφορά σε διαφορετικά επίπεδα. Εκεί τα πράγματα είναι περίπλοκα αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι το έργο της Επιτροπής που είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων και της εφαρμογής της ε, νομοθεσίας, άρα αναπόκειται σε εκείνους να επιταλέσουμε αυτό το έργο. Ε, φυσικά, εάν ε, υπάρξουν αυτοί οι πίνακες αντιστοίχησης, θα γίνει πιο εύκολη η ζωή τους. Αλλά είναι κάτι το αυτή τη στιγμή δεν είναι υποχρεωτικό και γι' αυτό θα ήθελα να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση από το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την ουσία. Όσον αφορά για το FFM, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη δυνατότητα να απαντήσω με λεπτομέρειες. Δεν είπα πάρα πολλά πράγματα στα εισαγωγικά μου σχόλια. Υπάρχουν το άρθρο 324 ε, το οποίο ε, προβλέπει την εμπλοκή του Προέδρου. Τακτικές συναντήσεις θα γίνουν μεταξύ Προέδρου του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, αυτό έγινε τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο, μια τέτοια συνάντηση και η επόμενη θα λάβει χώρα τον Απρίλιο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι πρόεδροι θα συζητήσουν ζητήματα προπολογισμού, κάτι το οποίο έγινε κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας. Επίσης, το ζήτημα του FFM, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και θα συζητηθεί στην αρχή της συνεδρίασης. Θα υπάρξουν λοιπόν αυτές τις τακτικές επαφές. Βεβαίως θα γίνουν κανονικές διαπραγματεύσεις. Ε, επίσης υπάρχει το άρθρο 312 το οποίο θα εφαρμοστεί υπό την εξή έννοια. Θα προτείνουμε οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου να έχουν μια ανταλλαγή απόψεων με την Προεδρία ε, την ε, επικείμενη Τρόικα πριν από κάθε συνεδρίαση εφόσον τίθεται στην μερίσια διάταξη το ζήτημα του FFM. Και αυτό δημιουργεί μια ευκαιρία για τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου να δώσουν τη δική τους συμβολή. Και στη συνέχεια η Προεδρία θα ενημερώσει τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου για την έκβαση αυτών των συναντήσεων και βεβαίως εγγυόμεθα μία πρόσβαση εκ μέρους του Κοινοβουλίου στα έγγραφα τα οποία, στα οποία βασίζονται οι συναντήσεις αυτές και αυτά τα οποία εκδίδονται μετά. Λοιπόν, έχουμε την υποστήριξη εδώ της ε, Τρόικα και έλαβε γνώση και η Κορεπέρ και νομίζω θα στηθεί σύντομα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία λοιπόν. Τώρα τι γίνεται με τους 18 ε, βουλευτές. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να επικυρώσουν το πρωτόκολλο σύμφωνα με τις απαιτήσει των εθνικών συνταγμάτων. Όσον αφορά την Ουγγαρία, ήδη αυτό έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο και προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία στην Κορεπέρ στι 13 Μαρτίου καλέσαμε τι χώρε μέλη να ρυστικοποιήσουν την επικυρώση το ταχύτερο δυνατό και κατά τη διάρκεια αυτών των έξι μηνών μπορώ να σα πω ότι τώρα είναι 21 μέλη τα οποία προχώρησαν στην επικύρωση. Δηλαδή υπάρχουν έξι χώρες οι οποίες ακόμα καθυστερούν. Τώρα, όσον αφορά το MFF και τους ε, πόρους, αυτό θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα δούμε τι θα περιληφθεί στην ε, πρόταση της Επιτροπής, ποια ακριβώς θα είναι η διατύπωση στο σχέδιο πρότασης και είμαι σίγουρη ότι το Συμβούλιο θα το συζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει επίσης την ε, δυνατότητα να συγκαλέψει μια διακοινοβουλευτική συνέλευση με την συμμετοχή και των εθνικών κοινοβούλων. Βεβαίως και ούτε να το πράξει και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα εθνικά κοινοβούλια επίσης είναι σημαντικά και βεβαίως έχουν ενισχυμένο ρόλο λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας και χρησιμοποιούν όλο και χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις σχέσεις αρμοδιότητες. Νομίζω λοιπόν θα συνεχίσουν τα εθνικά κοινοβούλια να, θα, ελέγχουν τα εθνικά κοινοβούλια τις εθνικές ε, κυβερνήσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος ε, Τασκόφσκι για τη σχέση ανάμεσα σε εναλλασσόμενες προεδρίες και στη μόνιμη προεδρία αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μου έθεσαν ε, και οι συνάδελφοι στην συνάντηση που είχαμε στη Βουδαπέστη στις αρχές Ιουνίου. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μας καθοδήγησε ήταν ο πλήρης σεβασμός των συνθήκων, οι συνθήκες και ο πλήρης σεβασμός τους. Δεν θελήσαμε να κάνουμε περισσότερα από τις συνθήκες, σεβαστήκαμε τις συνθήκες. Θα πρέπει να ρωτήσετε και τον κύριο Βάν ή εγώ νομίζω ότι είχαμε μια εξαιρετική πάντως συνεργασία. Ο κύριος Βαν μας άκουσε προσεκτικά, ήμασταν σε μόνιμη συνεργασία με την ομάδα του Βαν Ο Πρωθυπουργό με τον Ρομπάι είχαν μηνιαίες συναντήσεις, πολλές φορές και πιο συχνές. Συζητήσαμε μαζί τους όλα τα θέματα, είχε και κάποια αιτήματα προς την Προεδρία, ήθελα μια καλή προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήμασταν υπεύθυνοι για τη σωστή προετοιμασία Ήμασταν υπεύθυνοι για διάφορα θέματα όμως η μετανάστευση και η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική που είναι εν μέρη ε, ΚΕΠΑ αλλά και όχι μόνο ΚΕΠΑ και ε, σίγουρα το ΚΕΠΑ δεν ήταν δική μας ευθύνη βέβαια και δεν είχαμε σε καμία περίπτωση τη φιλοδοξία να αλλάξουμε εμεί το περιεχόμενο της συνθήκης. Ε, νομίζω ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος για μια καλή συνεργασία και μπορέσαμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γι' αυτό νομίζω ότι αν στοχεύσει κανείς πάρα πολύ ψηλά τότε μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα γιατί δεν διασφαλίζει τη συνεργασία των υπολείπων οργάνων. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθούν προβλήματα. Έχουμε αρκετά αυτή τη στιγμή στην Ένωση. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μας. Για τις δαπάνες για την ΚΕΠΑ που ήδη περνάει το θέμα ουσιαστικά στο θέμα της απαλλαγής, μας περνάει στο θέμα της απαλλαγής. Ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για αυτό το θέμα. ήμασταν παρόντες και στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Εμείς προτείναμε νέες λύσεις και νοτόμες για το θέμα της απαλλαγής. Το Κοινοβούλιο απέριψε την πρότασή μας τον μήνα Μάιο. Σέβομαι την άποψή σας, αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο θα επαναλαμβάνουμε τη συζήτηση για την απαλλαγή. Αν αυτό θέλει το Κοινοβούλιο, ε, έχει καλό, αλλά εμείς νομίζουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση για να πράγματι για να ξεμπερδεύουμε θα έλεγα σε εισαγωγικά με την απαλλαγή για κάποιους από το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο πάντως το θέμα παραμένει ανοιχτό και είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη λύση για τον κύριο Γκουαλτιέρη και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εγώ νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν έχει πράγματι όπως είπατε νομική βάση, αλλά δεν είναι ένα νομοθετικό κομμάτι μόνο, είναι στην ουσία ένα μέσο και ένα χρονοδιάγραμμα. Ήταν μια πολιτική απόφαση, πολύ σημαντική απόφαση, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη να γίνονται σεβαστές και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή που έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο να ελέγχουν αν οι υποχρεώσεις οι ανηλυμένες των κρατών μελών γίνονται αντικείμενο σεβασμού ιού. Συνεπώς λοιπόν η προσπάθεια ξεκίνησε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήθηκαν τα θέματα αυτά σε όλες τις μορφές των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να προωθήσουν τα προγράμματα σύγκλησης, τα προγράμματα τα μεταρρυθμιστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αξιολογήσει τις υποχρεώσεις αυτές. Αυτές οι αξιολογήσεις προκαλούν μερικές φορές κάποιες αντιτιθέμενες απαντήσεις, αλλά έτσι έχει η ζωή. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ανεξάρτητο σώμα προσπαθεί να κάνει ανεξάρτητες αξιολογήσεις των ε, πολιτικών των κρατών μελών. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στο ΕΚΟΦΗΝ την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο για να συζητηθούν όλα τα θέματα αυτά και οι αξιολογήσεις αυτές από την Επιτροπή, της Επιτροπής έτσι ώστε το πακέτο αυτό να περάσει για απόφαση στο Συμβούλιο. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν γι' αυτό σε αυτή τη φάση μια βάση στη συνθήκη. Έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική προσπάθεια σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε κάνει πριν από τη συνθήκη με την μέθοδο ανοιχτής συνεργασίας η οποία δεν ήταν και τόσο επιτυχή σαν μέθοδος. Περισσότερη διαφάνεια λοιπόν και ένα άλλο θέμα σχετικά με το λεγόμενο το εξαπλό πακέτο στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου θα ακουστεί ότι έχουν γίνει αρκετές υποχωρήσεις από το Συμβούλιο προς το Κοινοβούλιο για το πώς θα συμπεριλάβουμε και θα κάνουμε αναφορές περισσότερες στα πλαίσια του εξαπλού πακέτου στις θέσεις του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι έτσι και το Κοινοβούλιο θα βλέπει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και εξελίσσεται το ε, ε, ευρωπαϊκό εξάμεινο. για την εξωτερική εκπροσώπηση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα επηρεάσει νομίζω τη ζωή της κάθε Προεδρίας. Έχουμε εργαστεί σκληρά, όχι σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά κατά περίπτωση σε πολλές διεθνείς διασκέψεις τις οποίες πήραμε μέρος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Κάθε θέμα και κάθε συνάντηση είναι διαφορετική με διαφορετική νομική βάση. Η ΚΕΠΑ είναι κάπως πιο απλή αλλά εκεί υπάρχουν και πάρα πολλές μικτές αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια κάποια ερμηνεία, τα κράτη-μέλη μπορεί να δίνουν μια διαφορετική. Και γι' αυτό αυτό το οποίο εμείς κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε και να βαθιστούμε στις εμπειρίες των προηγούμενων διαπραγματεύσεων αλλά πάντα κατά περίπτωση. Και νομίζω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία που συμφωνήσαμε στα θέματα της, των δασών, της πολιτικής της δασικής, όπου υπήρχαν διαφορετικές απόψεις στα κράτη-μέλη, αλλά τώρα ξεκαθαρίστηκε λίγο το θέμα, ποιος θέλει τι, ακόμα και ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις αυτές σε κάποιες πρωτεύουσες, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη, κάποια θέματα πήγαν εύκολα, κάποια άλλα συζητήθηκαν με δυσκολίες. Παρόλα αυτά καταλήξαμε σε κάποια αποτελέσματα και μας συνεχάρισαν τα κράτη-μέλη την προηγούμενη εβδομάδα για τις λύσεις τις οποίες καταλήξαμε. Είναι σαφές ότι η συνθήκη εδώ δεν κάνει τη ζωή μας εύκολη γιατί δεν διευκρινίζεται σαφώς το ποιος κάνει τι Συμβούλιο, Κρατημέλη και Επιτροπή. Παραμένει λοιπόν το θέμα αυτός, ε, θα είναι ένας πονοκέφαλος και για τις επερχόμενες προεδρίες για τον κύριο Έφνερ για την πρωτοβουλία των πολιτών και τις υπογραφές ε, ενδικτύων. Εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και να προωθήσει την εμπλοκή των κρατών μελών. Υπάρχει ανάγκη για συνεργασία, αλλά αυτό είναι θέμα της Επιτροπής και όχι του Συμβουλίου. Και το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει το πώς θα προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Εσείς είσαστε τα αφεντικά στο συγκεκριμένο θέμα, συνεχίστε να τα ελέγχετε και στις 30 Ιουνίου θα έχουμε την πρώτη συνάντηση εμπειρογνωμόνων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να δώσω απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις οι οποίες μου τέθηκαν. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας και να αντισεβόμεθα πλήρως. Εκεί όπου η συνθήκη δεν είναι ξεκάθαρη, η ζωή μας περιεπλάκει. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Νομίζω ότι αν επιμείνουμε σε αυτήν την κατανομή εργασίας όπως προβλέπεται από τη συνθήκη και αν δεν ελέγχουμε συνεχώς τα όρια στα οποία, τα οποία αντιμετωπίζουμε ε, και ασχοληθούμε με την ουσία περισσότερο, τότε ίσως ε, να βρεθούμε σε καλύτερη, σε καλύτερη διάθεση, κάτι το οποίο θα βελτιώσει τις σχέσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας, είμαι θα ευγνώμονες, θεωρούμε ότι ο ρυθμός τον οποίο ακολούθησε η Ουγγαρία αυτό το εξάμεινο και το σύνθημά σας μια ισχυρή Ευρώπη με ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι ένα απλό σύνθημα αλλά είναι μια αρχή που θα ισχύει πάντα. Ευχαριστώ.